Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αρχίζουμε το δεύτερο κομμάτι των ακράσεων που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο των εργασιών μας για να συλλάβουμε σε γενικέ έννοιε αυτό που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπολογισμό της Ευρωζώνης η διακυβέρνηση της Ευρωζώνης δεν έχει ανταποκριθεί σε όλες τις προσδοκίες, κυρίως όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση και ασφαλώς υπάρχει περιθώριο πρόοδου. Έχουμε λοιπόν λάβει πρωτοβουλία μιας εκθέσεως με ακριβώς αυτό το θέμα, εκθέσεως σχετικής με την διακυβέρνηση και τον προϋπολογισμό της Ευρωζώνης. Ε, παρακολουθήσω μια σειρά από ε, παρεμβάσεις, από τοποθετήσεις ε, προερχόμενες από άτομα εκτός του Κοινοβουλίου που μας φώτισαν σε αυτό το θέμα αλλά βέβαια θέλουμε να ακούσουμε και άλλες προτάσεις. Ο Ρόμπερτο Γκουαλτιέρη καθώς οι δύο επιτροπές ΕΚΟΝ και ΜΠΑΤΣ Οικονομικών Νομισματικών Θεμάτων και Προϋπολογισμού είναι ε, στην αλλά ε, χρειάστηκε να αποχωρήσει, θα τον θα αντικατασταθεί. Ο κύριος Μπενουά Κεγέ, λοιπόν, συγκεκριμένος μας από την, ε, την Εκτελεστική Επιτροπή της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο κύριος Γκλάσνοκ από την Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων των Κάτω Χωρών και ο κύριος Σαβιές από την Οικονομική Σχολή Παρισίων. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Κεγέ εδώ θα αναφερθεί στο θέμα του ενός ευρωπαϊκού προϋπολογισμού χωρίς όμως να χρειάζεται να επεκτεθεί σε ιδιαίτερα στοιχεία μιας νομισματικής πολιτικής και έτσι κάποια στιγμή σας χρειαστεί ένα, όπως λέμε, policy mix οικονομικής και νομισματικής πολιτικής, δηλαδή μείγμα. Ο κύριος Καλής ασθενή και δυστυχώ δεν μπόρεσε να έρθει. Λοιπόν, δίνουμε πέντε λεπτά στον κάθε έναν από τους ηγητές καταρχάς για να κάνουν την ε, εισαγωγική τοποθέτηση για την ε, ακρόαση αυτή και μετά ομιλεί ο ένα και ε, αντίστροφα στο τέλος θα μιλήσουν δεύτερος αυτός που είχε μιλήσει πρώτος και Τούμπαλιν. Μετά ακούμε τους ε, ομιλητές μας, προσκεκλημένους μας, ε, στη συνέχεια πάλι τους ε, εισηγητές, τους και οδησηγητές, για δύο λεπτά τον καθέναν. Οι ειδικοί θα έχουν πέντε λεπτά για να δώσουν απαντήσεις στο σύνολο των ερωτήσεων που θα έχουν διατυπώσει και οδησηγητές και εάν μας μείνει χρόνος, αγαπητοί συνάδελφοι, μπορείτε να μιλήσετε εσείς για να κλείσουν οι δύο συνεισηγητές την συνεδρίαση και δίνω το λόγο στον κύριο Μπενουά Κυρέ. Τον ευχαριστώ που είναι εδώ παρόν και βέβαια μαζί στο πρόσωπό του ευχαριστώ όλους τους προσκεκριμένους μας. Αλλά λησμόνισα ότι πρώτα πρέπει να γίνει η παρουσίαση από τους Κυρία Μπερές, συμπαθάτε με. Βεβαίως και σας συγχωρώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τους προσκεκλημένους μας που είναι εδώ με το Ράιμερ Μπούγκε από τη στιγμή που αυτό το καθήκον. Έχουμε κατακλειστεί από πραγματογνωμοσύνες, ε, γνώσεις και εμπειρία σωρευμένη το 2012, πλουσιοτάτη. Αποφασίσαμε λοιπόν οι δύο επιτροπές μας να ξεκινήσουμε για πρώτη φορά με μια τέτοια έκθεση και είναι η πρώτη φορά νομίζω που το Κοινοβούλιο ε, αναφέρεται σε ένα θέμα το οποίο ειδικά αφορά την Ευρωζώνη, τον προπολογισμό της Ευρωζώνης. Θα μπορούσε μάλιστα να έχει προκύψει το θέμα, να προκύψει το θέμα αυτό την εποχή της συνθήκης του Μαστρίχτ. Αλλά τότε είχαν ε, ε, προβλεφθεί διαφορετικοί μηχανισμοί για να λειτουργήσει αυτό λειτουργήσανε μεν για ένα διάστημα, αλλά τελικά ήρθε η κρίση και έτσι αυτή η δημιουργική αβεβαιότητα της συνθήκης του Μαστρίχτ αποδείχθηκε τη σπάση ότι ήταν καταστροφική και αυτό αναγνωρίστηκε άλλωστε και από τις εργασίες του 2012, blueprint, ε, ε, τέσσερις έξι των τεσσάρων προέδρων και πριν από αυτό προτάσεις του Φαν Ρόμποη προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και μετά βλέπουμε λοιπόν τι υπάρχει εδώ επιτάπητος, περισσότερη ανάγκη λοιπόν για ε, εμπειρογνωμοσύνη, γνώσεις ε, κτλ. Γιατί δεν αν υπήρχε όλη αυτή η εμπειρογνωμοσύνη και οι γνώσεις δεν θα, αρκού, δεν θα παρά να ε, συνοψίσουμε τα υφιστάμενα δεδομένα ο Ράιμερ και εγώ. Δεν υπάρχουν όμως, οπότε πρέπει να δημιουργήσουμε νέο υλικό, να δώσουμε απαντήσεις, να σταθμίσουμε θέσεις διαφορετικές πολύ συχνά εγώ πολύ συχνά αρχίζω να βλέπω με έναν τρόπο πολύ πιο οργανωμένο το γιατί χρειάζεται ένας ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, ένας προϋπολογισμός της Ευρωζώνης, σημειώνω, ε, προσπαθώντας να είμαι στον τον πιο Ο πρώτος λοιπόν, η πρώτη λειτουργία θα ήταν σταθεροποιητική σε σχέση με συμμετρικές ε, ε, ασύμετρους κλειδονισμούς. Δεύτερη λειτουργία, διατήρηση δυνατοτήτων επενδύσεων πέραν των περιορισμών που μερικές φορές επιβάλλει το Σύμφωνο Σταθερότητας και βέβαια η διατήρηση της ε, σύγκλησης πέραν των μηχανισμών του προπολογισμού της Ένωσης που δεν έχουν αποδείξει αποτελεσματικότητα για την ε, σύγκληση στην Ευρωζώνη και αυτό το λέω επίοικος. Υπάρχουν διάφοροι τύποι πιθανών πόρων. Ε, πρώτον, μια εμβρυϊκή μορφή προπολογισμού της Ευρωζώνης με έναν Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και όλο το δυναμικό που μπορεί αυτός να έχει και όλο το, όλες τις δυνατότητες αξιοποίησης που θα μπορούσε κανείς να αναλογιστεί αν, αναλογ... σκεφτούμε κιόλα ότι τίθεται και το ζήτημα της ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης. Όλα αυτά είναι μέσα για την ε, απόκρουση συμμετρικών ή αντισυμμετρικών κλειδονισμών ε, που ε, χρειάζεται όσο δεν υπάρχουν αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί αντιστάθμισης όπως σε παραδείγματι ένα επίδομα ανεργίας ή κάτι αντίστοιχο. Στο θέμα της σύγκλησης και πέραν των περιορισμών που αμφισβητήθηκαν εκείς, και άλλων ε, διαρθρωτικών αναπροσαρμογών που μας έχουν απασχολήσει στο πλαίσιο του του δημοσιονομικού πλαισίου κτλ. θα μπορούσαν να είναι κάποιες ιδέες. Τούτων λεχθέντων, και δεν νομίζω να συγκλονίστηκε κανείς από αυτά που είπα, ε, αυτό που δεν βλέπουμε ο Ράιλερ και εγώ είναι ε, πού θα αναστήσουμε τα καλά εκείνα ε, επιχειρήματα ώστε να πείσουμε τους αρμόδιους για τη λήψη των αποφάσεων. Οι οποίοι σήμερα ποιοι είναι, είναι αυτοί οι οποίοι πολύ συχνά συνεδριάζονται στο Eurogroup, στο ECOFIN ή κυρίως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβαν αποφάσεις. Η δική σας λοιπόν συμβολή σήμερα θα μπορούσε να μας προσφέρει ε, ιδέες πρώτα απ' όλα για το ποιες θα ήταν οι καλύτερες λύσεις αλλά και περισσότερο ποια θα ήταν τα καλύτερα επιχειρήματα για να πούμε όχι ε, ε, εάν πρέπει να κάνουμε αυτό το επιπλέον βήμα, αλλά πώς θα πείσουμε αυτούς που πρέπει να λάβουν τη σχετική απόφαση. Ευχαριστώ, Περβόνς. Κύριε Μπέο, εσείς θα κλείσετε, έτσι. Κύριε Κερέ, έτσι το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, Θα μιλήσω αγγλικά, αλλά θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τους δύο πρόεδρους των Επιτροπών και τους δύο εισηγητές για την οργάνωση αυτής της ανταλλαγής απόψεων, προκειμένου να προωθηθεί η δημόσια συζήτηση για τη δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης και μάλιστα ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ένα σημαντικό πολιτικό βήμα. Και θα αναφερθώ στην ανάγκη αυτής της πολιτικής προσέγγισης, κάτι που ε, σχετικοποιεί αυτά που θα σα πω ως ε, κεντρικό τραπεζίτη, γιατί δεν έχω πολιτικό κύριο. Παίρνω στα αγγλικά τώρα. Όλοι γνωρίζουμε ότι η πολιτική προσοχή είναι εστιασμένη αλλού αυτή τη στιγμή, κάτι που δεν είναι λόγος για να ξεχνούμε το στόχο τη ολοκλήρωση του ΟΝΕ, τη ναι, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, δηλαδή θωράκιση τη ανθεκτικότητα τη ΟΝΕ ναι, για να μπορεί να απορροφά του κραδασμού και επίση να δημιουργήσει οικονομική εμπιστοσύνη για να τονώσει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Παρόλο που η πολιτική προσοχή ε, περισπάται προς άλλες κατευθύνσεις αυτή τη στιγμή. Ε, και φυσικά, αν υλοποιηθούν οι κίνδυνοι ε, της χαμηλής ανάκαμψης δεν θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε ούτε την προσφυγική κρίση ούτε να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Ας το έχουμε και αυτό υπόψη. Μία σύντομη ματιά στι ε, δημοσιονομικέ πολιτικέ σήμερα μα πείθουν για την σημασία αυτή τη συζήτηση σήμερα. Γιατί η ανάκαμψη στην Ευρωζώνη ε, ακολουθεί χαμηλού ρυθμού, κυρίω στηρίζεται από τα νομισματικά μέτρα της ΕΚΤ και τη χαμηλή τιμή των ενεργειακών προϊόντων. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε ε, γεωπολιτικούς κινδύνους και αυξανόμενη αβεβαιότητα. Και πολλές χώρες εξακολουθούν να βρίσκονται σε μια πολύ ευάλωτη κατάσταση. Μάλιστα αυτή η κατάσταση δημιουργεί αφιβολίε για την, αντιμετώπιση, ε, για την ικανότητα της Ευρωζώνης να αντιμετωπίσει μελλοντικού οικονομικούς κραδασμού. Θα πρέπει λοιπόν να διασκεδάσουμε αυτέ τις αμφιβολίες σήμερα και να θωρακίσουμε την Ευρωζώνη για τους μελλοντικού ε, κινδύνους. Και μάλιστα ως μέλος τη κεντρική Τράπεζα, ε, δεν πρόκειται να σα εξηγήσω εγώ ποια θα ήταν η κατάλληλη δημοσιονομική ικανότητα για την Ευρωζώνη. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή που θα απορρεύσει από μια πολιτική συζήτηση. Εγώ θα σα κάνω μια εκτίμηση για το, τι, για το γιατί χρειαζόμαστε μια δημοσιονομική ικανότητα και γιατί δεν είναι βέβαια η πανάκια που θα κάνει την ΟΝΕ ναι καλύτερη. Αλλά θα πρέπει να δούμε υπό ποιου όρου θα μπορούσε να λειτουργήσει. Η Ευρωζώνη σήμερα δεν βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι ε, μεταξύ ε, αντίθετων κατευθύνσεων αφενός δηλαδή τις υπεύθυνε δημοσιονομικές πολιτικές και την, και την άλλη κατεύθυνση την, κοινή, την δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιλογή στηρίζεται σε ιδεολογικούς και πολιτικούς ρόλους, αλλά από οικονομική άποψη δεν υπάρχει καμία διάσταση κατευθύνσεων. Είναι αλληλοσυμπληρούμενες. Προπόθεση για να μπορούν οι δημοσιονομικέ πολιτικέ να συμβάλλουν στη μακροοικονομική σταθεροποίηση είναι να εξασφαλίσουν ότι οι χρηματοπιστωτικέ αγορέ και οι πολίτε έχουν εμπιστοσύνη στη βιωσιμότητα των οικονομικών πολιτικών. Γι' αυτό είναι σημαντική αυτή η βιωσιμότητα. Δεν είναι θέμα θεολογικό-ιδεολογικό, είναι οικονομικό και πολιτικό και είναι επιτακτική ανάγκη Θέλουμε να έχουμε ε, εμπιστοσύνη στη διακυβέρνηση για, την, ε, για το συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών και θα πρέπει και οι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη ε, ότι τηρούνται οι κοινοί κανόνες. Οποιαδήποτε κοινή δημοσιονομική ικανότητα θα, θα χρηματοδοτείται είτε από εφιστάμενους είτε από μελλοντικού φόρους των ίδιων φορολογουμένων, από τους ίδιους φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν τους Εθνικού προπολογισμού. Οπότε, αν δεν έχουμε υγιεί ε, εθνικού ε, προπολογισμού, δεν θα έχουμε ε, γερά θεμέλια για να δημιουργήσουμε και μια τέτοια κοινή δημοσιονομική ικανότητα. Οπότε τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ξαναφτιάξουν τέτοιους ε, προφυλακτήρες ε, εθνικούς για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τους μελλοντικού ε, κραδασμούς. Τώρα, γιατί χρειάζεται μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και ανάπτυξη, της ανανέωση ή της συμπλήρωσής του για να γίνει πιο αποτελεσματική, να αυξηθεί η συμμετοχή των κρατών μελών, να κάνουν κτήμα του. και πρόκειται για διακλαδώσει που ξεπερνούν την σημερινή συζήτηση, εύλογη συζήτηση, αλλά ανήκει σε διαφορετικό επίπεδο σε διαφορετική ευκαιρία. Και αν θα αρχίσουμε να ξυλώνουμε τους υπάρχοντες κανόνες δεν πρόκειται να δημιουργήσουμε ε, εμπιστοσύνη, την ενισχύσουμε. Πρώτα πρέπει να εφαρμόζουμε τους υφιστάμενους κανόνες. Επίσης, χωρίς ε, εργαλεία νομισματικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, αυτή είναι ο ορισμός της νομισματικής ένωσης, η δημοσιονομική πολιτική θα παρεμποδιστεί αν ε, η κραδασμοί είναι πολύ σοβαροί και δεν υπάρχει απορρόφηση, δυνατότητα της οικονομίας να απορροφήσει αυτού τους κραδασμούς, η δυνατότητα του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Οπότε θα πρέπει να μειώσουμε το μέγεθος αυτού του κραδασμών. Γι' αυτό κάνουμε και την Τραπεζική Ένωση. Να μειώσουμε την πιθανότητα ή το μέγεθος ε, ισχυρών ε, οικονομικών κραδασμών. Και αυτό αυτή την πορεία ακολουθεί η Τραπεζική Ένωση. Όμω δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι από εδώ και πέρα η Ευρωζώνη θα είναι στο απειρόβλητο των κρίσεων. Γι' αυτό και ζητήσαμε να ενισχυθεί η δυνατότητα απορρόφηση κρατοσμών σε επίπεδο Ευρωζώνη και να συμπληρωθούν οι σταθεροποιητέ ε, που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο. Τώρα, πώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δημοσιονομική ικανότητα μπορεί να έχει τη μορφή, ε, τη μορφή μακροασφάλισης, ε, ασφάλισης ενεργείας ε, ή εξασφάλιση δημοσίων αγαθών. Η επιλογή σε τελική ανάλυση είναι πολιτικού χαρακτήρα, είναι πολιτική απόφαση, αλλά είναι ευκαιρία να έχουμε μια συζήτηση για τους συλλογικούς στόχους στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη. Και αυτή η συζήτηση είναι χρησιμότερη από ποτέ και ξεπερνάει το οικονομικό επίπεδο. Δεν πρόκειται να επισέλθω σε υπερβολικέ λεπτομέρειε. Πάντω πιστεύω ακράδαντα ότι η συζήτηση είναι κυρίω πολιτική και δεν μπορούμε να βοηθήσουμε εμεί ε, ω κυβέρνητε ε, μέλη τη ΕΚΤ. Θα πρέπει να μεγιστοποιήσουμε πάντω τα θετικά αποτελέσματα τη λειτουργία τη Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Και εδώ θα πρέπει να διαπιστώσουμε πρόοδο σε τρει διαστάσει. Πρώτη διάσταση είναι η συγκέντρωση των δημοσιονομικών πόρων άσχετα της φύσης τους, του μεγέθους τους. Αυτό θα ισχύσει και θα λειτουργήσει μόνο αν η αλληλεγγύη ε, συμβαδίζει με την υπευθυνότητα. Δηλαδή να έχουμε, για να έχουμε μια δημοσιονομικό επιμερισμό των ευθυνών στην Ευρωπαϊκή, στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, θα πρέπει να έχουμε κοινέ διαδικασίες λήψης αποφάσεων με ισχυρά κοινά θεσμικά όργανα για να είμαστε αποτελεσματικοί και μια πρόσβαση στην κοινή δημοσιονομική ικανότητα θα πρέπει να εξαρτάται από τη συμμόρφωση των κριτηρίων του Συμφώνου σταθερότητα και Ανάπτυξης. Επίσης, στόχο μας είναι να ε, μην επιβαρύνουμε τις δημοσιονομικές πολιτικές ε, και να διευκολύνουμε την ε, μακροπροσαρμογή. Δηλαδή θέλουμε όσο περισσότερη δημοσιονομική ικανότητα χρειάζεται, αλλά όσο, όσο περισσότεροι και οι μηχανισμοί αγοράς χρειάζονται. Επίσης θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την τραπεζική και την, και κεφαλαία αγορά μάλιστα και να ενισχύσουμε την αφεκτικότητα της Ευρωζώνης και επίσης να ολοκληρώσουμε και την ενιαία αγορά συμπεριλαμβάνοντας και την ενιαία αγορά των υπηρεσιών. Έτσι, ε, να περιοριστεί ο, η ανάλυση του κινδύνου από το δημόσιο τομέα. Κατά τη γνώμη μου, στην καρδιά της αρχής της ασφάλισης είναι η εκ των προτέρων κατανομή των κινδύνων. Οπότε οποιαδήποτε κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να συνοδεύεται από μια διαδικασία σύγκλησης προς πιο ανθεκτικές οικονομίες. Χρειαζόμαστε ένα καθαρό δρόμο μεταρρυθμίσεων και μια διαδικασία σύγκλησης που θα κάνει τις οικονομίες από κοινού πιο ανθεκτικές στους κραδασμούς. Και φυσικά απαιτείται και οικονομική σύγκληση. Γιατί αν θέλετε μια νέα διαδικασία οικονομικής σύγκλησης, θα πρέπει να επανεφεύρετε κάποιε αρχέ να συμφωνήσετε στους μηχανισμούς και να κάτι τέτοιο και μια πολιτική σύγκληση. Και εν κατακλείδη, η προστασία κατά των μικρών κινδύνων, ε, κατά του ηθικού κινδύνου, συγγνώμη, που βρίσκεται στο επίκεντρο τη συζήτηση, είναι σημαντική, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω στρατηγική για για να αναβάλουμε επαόριστον τη, δημοσιονομική ικανότητα. Αν θέλουμε μια δημοσιονομική ικανότητα θα πρέπει να το κάνουμε προοδευτικά, υπό όρους, υπό προϋποθέσεις και να συμβαδίζει με την επαναφορά δημοσιονομικών buffer σε εθνικό επίπεδο, ε, επαναφορά της δημοσιονομικής ικανότητας σε εθνικό επίπεδο, δυνατότητα σύγκλησης ε, σε εθνικό επίπεδο για την απορρόφηση κινδύνων και ενίσχυση των θεσμικών οργάνων σε επίπεδο ευρωζώνης, ώστε να έχουμε ισχυρούς κοινούς θεσμούς που να μπορούν να λειτουργούν σε αυτή την κοινή δημοσιονομική ικανότητα. Ολοκληρώνω λοιπόν. Εδώ βάζω τελεία, γιατί θα μπορούσα να μιλάω για πολλή ώρα. Χαίρομαι πάντως που κηρύξατε το εναρκτήριο λάκτισμα αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρουσίαση κύριε Κερέ για το φω που ρίξατε στην υπόθεση. Και βλέπουμε ότι χρειάζεται και πολιτική στράτευση για ένα τέτοιο εγχείρημα. Θα δώσω τώρα το λόγο στον ε, διευθυντή της Κεντρικής Τραπέζας ε, των Κατοχωρών, στον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας των Κατοχωρών, τον κύριο Κνότ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Εισηγήτρια, κύριε Εισηγητά, μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να συμμετάσχω σε αυτή τη δημόσια ακρόαση για την δημοσιονομική δυνατότητα της Ευρωζώνης και να παρουσιάσω και τις απόψεις μου στο Ευρωκοινοβούλιο. Ελπίζω να σας διευκολύνουν στην μελέτη του θέματος που σα απασχολεί. Ήδη νομίζω το έγγραφο που σας μοιράστηκε είναι μια προσέγγιση ποικίλη για τις προοπτικές μιας δημοσιονομικής δυνατότητας. Τι θα μπορούσε να πετύχει και τι όχι έχει μια οπτική γωνία αρκετά ευρεία με πολλές ενδεχόμενες λειτουργίες αυτής της δημοσιονομικής οργάνωσης όπως την σύγκληση, την κινητοποίηση για μεταρρυθμίσεις και τον δανειστή έσχα λύση. λύσης. Ε, σήμερα θα ήθελα να επικεντρωθώ στην σταθεροποίηση και την αντιμετώπιση των συμμετρικών κινδύνων, δηλαδή το πλέον ε, το πλέον σημαντικό στοιχείο με προστιθέμενη αξία. Για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Σταθεροποίηση ήθελα να μιλήσω λοιπόν για τον αντίκτυπο που μπορεί να προκληθούν από του αντίξου οικονομικού κύκλου και το πώς όλα αυτά μπορεί να επιδράσουν στην Ευρωζώνη και σε επίπεδο κρατών μελών. Για τη διαφορά μεταξύ της κατανομής κινδύνου εξάντε και την κατανομή εξ, εξ, ε, τη μια την άλλη κατεύθυνση και επίση για τη σημασία τη κατανομή κινδύνου μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Πριν περάσω σε όλε αυτέ τι λεπτομέρειε, πρώτα απ' όλα μια επισκόπηση του πώ νομίζω ότι θα πρέπει να διοργανωθούμε δημοσιονομικά κατά τη διάρκεια τη κρίση. Στην αρχή ο ομοσπονδιακό προπολογισμό για την Ευρωζώνη δεν φαινόταν απαραίτητο, διότι φαινόταν ότι οι ασυμμετρικοί κινδύνοι μπορούν να αντιμετωπιστούν από τι χώρε από του εθνικού του προπολογισμού, αρκεί να ακολουθούσαν το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Δυστυχώ η κατάσταση απέδειξε ότι αυτό δεν ίσχυε και πολλέ χώρε με τι δημοσιονομικέ του πολιτικέ δεν μπόρεσαν να ε, αξιοποιήσουν τι δυνατότητε σταθεροποίηση. Αυτό οφειλόταν εν μέρη στην, μη, ε, ε, στην πλημελή πειθαρχία και σε σεβασμό των στόχων του συμφώνου. Κάποιες χώρες είχαν ε, σωστά δημοσιονομικά ή έστω ένα σχετικό έλλειμμα μόνο θεωρητικά και ποτέ στην πράξη. Έτσι, ο αντίκτυπο τη κρίση ε, πολλαπλασιάστηκε από τι πολλέ μακροοικονομικέ ανισορροπίε που είχαν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Οι χώρε που είχαν, είχαν τι περισσότερα σοβαρέ ανισορροπίε, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Ισπανία, με έλλειμμα στον προπολογισμό το 2009 κατά μέσο όρο 11%, 11 μονάδε του ΑΕΠ, παραπάνω από ό,τι προβλεπόταν την περασμένη χρονιά. Ε, το διπλάσιο τουλάχιστον. Ε, έτσι, η δημοσιονομική εξυγένση ήταν απαραίτητη για τα περισσότερα κράτη-μέλη και έτσι από το 2011 2014 η δημοσιονομική ε, τάση της Ευρωζώνης όδευε προς την συρρήκνωση. Ιδίω όταν φτάσαμε στα κατώτατα όρια τη ε, δημοσιονομική διοργάνωση. Σε αυτέ τι έκτατε συνθήκε, το Ταμείο Σταθεροποίηση ε, των Δημοσιονομικών θα μπορούσε να μα αντιμετωπι... βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε του ασυμμετρικού κινδύνου σε επίπεδο κρατών μελών και να υπάρχει ένα πιο ισόρροπο μείγμα πολιτικών για όλη την Ευρωζώνη. Ήταν βέβαια σαφέ πριν από την έναρξη τη Οικονομική και Νομισματική Ένωση ότι η σταθεροποίηση θα ήταν πολύ πιο δύσκολη στην πράξη από ό,τι στη θεωρία. Είναι δύσκολο να ε, βρεθούν οι όροι ώστε ένα τέτοιο ταμείο να είναι ε, αποδεκτό και από πολιτική άποψη, έτσι όπω έχει περιγραφεί στην έκθεση των πέντε Προέδρων. Πάντω, ε, εφόσον δεν υπάρχει ομοσπονδιακό προπολογισμό, το ταμείο αυτό θα πρέπει να είναι σχετικά μικρή κλίμακα και φαίνεται ότι θα είναι πολύ προβληματικό να μην υπάρχουν μεταφορέ ή να μην ε, επηρεαστεί από τι αρνητικέ τάσει στη δημοσιονομική πειθαρχία. Τρει πρακτικέ δυσκολίε λοιπόν και μια εναλλακτική. Αυτά ήθελα να τονίσω. Πρώτη, ε, δυσκολία και πρόκληση είναι ότι το είδος ασυμμετρικών διακυμάνσεων που είδαμε στην Ευρωζώνη είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν ε, αποτελεσματικά με περιορισμένες δημοσιονομικές δυνατότητες. Τα ταμεία σταθερότητας συνήθως αφορούν τους επιχειρηματικούς κύκλους, οι οποίοι έχουν μια διάρκεια περίπου οκταετία συνήθως. Ε, ένα, μια τέτοια περιορισμένη διάρκεια θα κάνει και τις συνεισφορές προς το Ταμείο ή τις κινήσεις από αυτό σχετικά προσωρινού χαρακτήρα. Αν όμως δει κανείς τα κάτι μέλη των, της Ευρωζώνης και τους επαγγελματικούς τους κύκλους είναι συγχρονισμένα κατά τρόπο αρκετά πρωτότυπο από το 2009. Οι ασυμμετρικές δικημάνσεις όμως στις διφρονομικές τους ε, διοργανώσεις είναι πολύ ε, πιο αποκλίνουσες και μακροχρόνιες, με διαφορετικούς δυναμικούς κύκλους που έχουν τουλάχιστον διπλάσια διάρκεια από τους επιχειρηματικούς κύκλους, 16 20 χρόνια. Αυτές οι ανισορροπίες συμπίπτουν και με τις εμένουσες αποκλήσεις την ανταγωνιστικότητα, στους τρέχοντες λογαριασμούς και στις τιμές της στέγης και των ε, προϊόντων. Έτσι, οι τελευταίες διακυμάνσεις ε, δοκίμασαν την κατάσταση στην πράξη, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαν ε, μελετηθεί αρκετά ούτε στην εκδοχή των πέντε πρόεδρων ούτε αλλού. Έτσι λοιπόν το Ταμείο που είχε λάβει υπόψη του μόνο τη διάρκεια των επιχειρηματικών κύκλων μπόρεσε να ε, σταθεροποιήσει μόνο ένα μέρο, να αντιμετωπίσει μόνο ένα μέρο του ευρύτερου δημοσιονομικού κύκλου. Όμω χρειάζεται πολύ πιο μακροχρόνιο προγραμματισμό με μεταφορέ και κινήσει ε, από ό,τι έχει ως τώρα προβλεφθεί. Η δεύτερη δυσκολία στην πράξη είναι ότι η δημοσιονομική δυνατότητα ε, αναπόφευκτα θα επηρεάσει τις εθνικές πολιτικές των, δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών μελών. Πρώτα απ' όλα μπορεί να αυξηθούν οι φόροι που ε, συλλέγονται σε, συγκεντρώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά πάντοτε μιλάμε για του ίδιου φορολογούμενου, του Ευρωπαίου πολίτε. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε να φορολογούμε του εξωγήνου από διάστημα. Ε, ε, ένα ομοσπονδιακό λοιπόν ε, ταμείο, μια ομοσπονδιακή διοργάνωση και προπολογισμό θα επηρεάζει και την εθνική φορολογία καθώς και το φορολογικό περιθώριο που διαθέτουν τα επιμέρους κράτη-μέλη. Αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να γίνει ακόμη πιο περίπλοκο εάν το ταμείο αυτό μπορούσε να δανειστεί για να καλύψει τους ελληματικούς αγοραστές στο ομοσπονδιακό και όχι μόνο στο εθνικό επίπεδο. Δεδομένων όμω των τωρινών επίπεδων φορολογία στα περισσοτερα τη κράτη-μέλη τη Ευρωζώνη, ένα τέτοιο ταμείο σταθεροποίηση και σταθερότητα δεν θα έπρεπε να οδηγήσει σε υψηλότερη φορολογία και δανεισμό. Αυτό σημαίνει όμω ότι το Ταμείο θα μπορούσε να επηρεάσει την επιβολή του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη και φαίνεται ότι η έκβαση αυτής της αναπόφευτης κίνησης προς την δημοσιονομική δυνατότητα σε επίπεδο ευρωζώνης θα έπρεπε να συμβαδίσει στενά με αυστηρότατη επιβολή των δημοσιονομικών κανόνων σε επίπεδο κατών μελών με μεγαλύτερη έμφαση στα επίπεδα του χρέους και τους έμεσους μελλοντικούς φόρους, καθώς και τα στοιχεία παθητικού που μπορεί να προκύψουν από αυτά. Η τρίτη δυσκολία στην πράξη είναι ότι το Ταμείο Σταθερότητας μπορεί να προκαλούσε και μεγαλύτερη δημόσια κατανομή κινδύνου, ε, μεταξύ των κρατών δηλαδή, που είναι και ο στόχος. Στην ευρωπαϊκή οικονομική και νομισματική πολιτική. Αυτή η κατανομή έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια κατά τρόπο αρκετά ε, θετικό. Όπω με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομική Σταθερότητα. Όμω το πρόβλημα που υπάρχει εδώ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση δεν λειτουργεί ακόμη ε, παρκώ σε κάποιου σημαντικού τομεί πολιτική. Τα κράτη-μέλη έχουν ακόμη σοβαρέ αποκλήσει και διαφέρουν όχι μόνο προ το δημόσιο χρέο ή τα ε, ισοζύγια πληρωμών, αλλά και ω προ την δυνατότητα προσαρμογή, την συνολική του δυνατότητα ανταγωνιστικότητα και τη θεσμική του ε, ευεξία. Εδώ λοιπόν ένα ταμείο σταθερότητα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κατεύθυνση μόνο μόνιμε μεταφορέ από μια, σε μια δίκαιη κατανομή κινδύνου που θα είχε προβλεφθεί εκ των προτέρων. Δηλαδή δεν έχει κανεί ιδέα εκ των προτέρων πού θα πρέπει να οδεύσουν οι πληρωμέ για την εξηγήση και τη διάσωση. Έπειτα, η περισσότερη κατανομή κινδύνου θα πρέπει να συνοδεύεται, κατά την άποψή μου, από πολύ περισσότερο πολιτικό συντονισμό και πολύ εντονότερε προσπάθειε για την ε, αναχέτηση του κινδύνου. Ε, θα πρέπει να υπάρχει ε, αυστηρότερο σεβασμό και του Συμφώνου Σταθερότητα και ανάπτυξη αλλά και των μακροοικονομικών ε, ανισορροπιών και τη διαδικασία αντιμετώπιση του, ώστε να αντιμετωπιστεί εκ των προτέρων η μετάδοση των μακροοικονομικών αυτών αποκλήσεων, προκαλώντα του τριγμού και του κλειδονισμού που είδαμε τα τελευταία χρόνια. Επίση, πρέπει να συνισχυθούν οι διάφορε δημοσιονομικέ δομέ, δηλαδή ένα πιο συντονισμένο τρόπο για την μεταρρύθμιση τη αγορά εργασία, λόγου χάρη. Έτσι, οι πολιτικοί ηθήνοντε θα πρέπει να σκεφτούν πολύ προσεκτικά το σχεδιασμό οποιοδήποτε κεντρικού μηχανισμού και των προποθέσεων για να υπάρξει σύγκληση σε όλου του πολιτικού τομεί τη Ευρωζώνη. Και εντωμεταξύ, τέταρτη και τελευταία παρατήρηση, ε, άλλοι τρόποι για να έχουμε περισσότερη ε, και καλύτερη αναχέτηση των κινδύνων είναι ε, να κοιτάξουμε τη μελέτη που δείχνει ότι για τις Ηνωμένε Πολιτείες ε, η κατανομή κινδύνου με τον ιδιωτικό τομέα, με τις ε, ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές αγορές, είναι ένα πολύ μεγαλύτερο και σημαντικότερο ποσοστό αντιμετώπιση των ασυμμετρικών κινδύνων, 62% δηλαδή, από ότι η κατανομή του κινδύνου μέσω του δημόσιου αποθεματικού που φτάνει το 13% με τον ομοσπονδιακό προπολογισμό. Άλλε μελέτε για τη Γερμανία και τον Καναδά δείχνουν ακριβώ τα ίδια αποτελέσματα. Η κατανομή κινδύνου λοιπόν με τον ιδιωτικό τομέα είναι ίσως και έχει μάλλον και περισσότερο δυναμικό από ότι σε κρατικό επίπεδο. Αλλά δυστυχώ έχει προωθηθεί πολύ λιγότερο στου ε, οικονομικού κύκλου. Οι ροέ των ιδιωτικών κεφάλων, κεφαλαίων μπορεί μάλιστα να έχουν οξύνει του κλειδονισμού και του τριγμού ε, σε ε, καιρού κρίση στα διάφορα κατημέλη με διαρροή κεφαλαίων. Πρέπει λοιπόν να έχουμε πιο εύρωστου τρόπου οικονομική και να προλάβουμε τις προκυκλικές διαρροές κεφαλαίων. Νομίζω ότι η Ένωση Χρηματαγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα, μια εξαιρετική ιδέα και πριν στραφούμε σε έναν ομοσπονδιακό προπολογισμό, το να αμβλύνουμε τους, ε, τα πλήγματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και να φροντίσουμε να αναχαιθήσουμε τον κίνδυνο είναι ήδη κάτι που μπορούμε να πετύχουμε σε επίπεδο αγορά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριος Ξαβιέ από το Paris School of Economics. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ τους συγγητές που μου δίνουν την ευκαιρία να εκφραστώ στο θέμα αυτό και τι θα τοποθετηθώ με προσωπικές μου απόψεις, εκπροσωπώ εδώ το οικονομικό παρατηρητήριο της Γαλλίας και τις διάφορες εργασίες που έχουμε κάνει, οικονομική ανάλυση για το θέμα το δημοσιονομικό της Ευρώπης. Θα μιλήσω γαλλικά με την αδειά σας. Θα πρέπει νομίζω να ξεκινήσουμε από μια σχετική διαπίστωση για να μιλήσουμε για την απόλυτη αυτή ανάγκη για τον προπολογισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια πραγματιστική προσέγγιση της οικονομικής συζήτησης που οδηγεί σε αυτή τη ε, συζήτηση για τη σταθεροποίηση που προβάλλουν στην εκθεσή τους πέντε πρόεδροι, πολύ εύστοχα, ένα κεντρικό καθήκον και νοφανές στον ε, Δημόσιο Ευρωπαϊκό Διάλογο σχέση με άλλες αποστολές που ανέφερε η κυρία Μπερές. Κεντρική σημασία πάντως ε, και που εξηγεί την εξέλιξη των συζητήσεων. Ένα άλλο θέμα που θέλω να προβάλλω σε αυτή την απόπειρα για προβολή επιχειρημάτων και πέραν του τεχνικού χαρακτήρα και των αναλύσεων που έχουν προβληθεί σε όλα αυτά τα θέματα του ευρωπαϊκού προπολογισμού, είναι ένας πραγματισμός, ρεαλισμός που ουσιαστικά συγκρίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλες ε, δημοσιονομικές ε, ομοσπονδίες, Καναδά, Πολιτείες, με συγκρίσιμα στοιχεία. Δηλαδή να κοιτάξουμε τι μπορεί ως σταθεροποίηση να φέρει αποτελέσματα και, και τι δεν δίνει σταθεροποιητικά αποτελέσματα. Και τρίτον, ε, πιο συγκεκριμένα εργαλεία στο πλαίσιο των ε, πολιτικών ορίων που εξετέθησαν και κυρίως την ιδέα της, ε, ενός ευρωπαϊκού, μιας ευρωπαϊκής ασφάλισης Θα μπορούσαμε λοιπόν να συμφωνήσουμε ότι από το μάθηση του Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης οι λύσεις που προτάθηκαν δεν μπόρεσαν να αντέξουν τους κλειδονισμούς μιας κρίσης διαστάσεων που δεν είχαν προβλεφθεί, δηλαδή που οδήγησαν σε ένα μεγάλο οικονομικό κλειδονισμό. Η ιδέα δηλαδή του Μαστρίχ που ήταν η νομισματική ε, πολιτική να έχει τη διαχείριση του κύκλου εξωτερώθηκε από τα μηδενικά επιτόκια, από την απουσία περιθωρίου χειρισμού ενός δημοσιονομικού εργαλείου για τα κράτη και από μια ζήτηση στις νευροζώνη πολύ χαμηλή, με πληθωρισμό πολύ χαμηλότερο από τους στόχους και με ε, χάσματα ζήτησης ε, σε ορισμένες χώρες σημαντικά. Πάνω απ' όλα με ασυμμετρίες μεταξύ των χωρών. Υπήρξαν λοιπόν διάφορες εξελίξεις στα ευρωπαϊκά κείμενα και ε, όροι ευελιξίας που εισήχθησαν αλλά ταυτόχρονα είτε πρόκειται για όρους ευελιξίας ή για μακροοικονομικές αναλύσεις, τα κείμενα αυτά καθιστούν πολύ δυσνόητη την ε, ανάγνωση των ευρωπαϊκών κειμένων, ακόμα και για οικονομικούς ειδικού εκτός των ευρωπαϊκών οργάνων και βέβαια την τήρηση των κανόνων, όπως αναφέρθηκε κοινότερα, γιατί πια δεν ξέρουμε ποιος κανόνας ισχύει όταν προσπαθούμε να διαγνώσουμε τη δυναμική της κάθε χώρας. Άρα λοιπόν πρέπει να διευκρινιστούν οι κανόνες, και να ε, επανέλθουμε στον αρχικό στόχο αυτόν που απέτυχε να ικανοποιήσει το μεθετόρα δόμημα τη σταθεροποίηση, μακροοικονομική σταθεροποίηση σε επίπεδο ε, και άρα αυτή την σταθεροποίηση πρέπει να την επιδιώξουμε με δεδομένη αυτή την, ε, δεδομένο το έλλειμμα ζήτησης. Για τις λοιπές λοιπόν δημοσιονομικές ομοσπονδίες ή νομισματικές ενώσεις μπορούμε να κάνουμε ως σύγκριση τον ελάχιστο προϋπολογισμό, γελία μικρό προϋπολογισμό της Ευρωζώνης σε σχέση με τις εισφορές των κρατών σε ποσοστό δαπανών ο, δι, ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός είναι 2% των δαπανών στην Ευρωζώνη, όχι των εισόδων των δαπανών, 2%. Στο δε Καναδά, που είναι το πιο αποκεντρωμένο συγκρινόμενο κράτος, είναι 8 πλάσια αυτά τα ε, ποσοστά για τις δαπάνες. Δεν υπάρχει δηλαδή δημοσιονομική ε, νομισματική ένωση που να λειτουργεί με τόσο χαμηλό προϋπολογισμό και να μπορεί να εξασφαλίσει νομισματική ένωση. Και έτσι φτάνουμε στη συζήτηση, στο κλειδί αυτή τη συζήτηση για την ε, σταθεροποίηση, που είναι ο συντονισμό πρώτα των εθνικών προπολογισμών, πρώτον, και δεύτερον, η χρήση συγκεκριμένων αντικυκλικών δημοσιονομικών εργαλείων επιπλέον αυτού του συντονισμού. Και βέβαια υπάρχει και το πρόσθετο ζήτημα που θα θέλαμε να εισαγάγουμε είναι και τα δημοσιονομικά εργαλεία βεβαίως να υπενθυμίσουμε αλλά και η αναζήτηση ομοσπονδιακών εργαλείων. Ο συντονισμό λοιπόν των δημοσιονομικών μέσων ή εργαλείων που θα μπορούσαμε να προτείνουμε πρέπει να διαρθρωθεί με μια ανάλυση οικονομική που θα καθιστούσε δυνατή την σύνθεση ενός Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, European Fiscal Board, που προτείνει και η έκθεση των πέντε προέδρων, ενός Δημοσιονομικού Συμβουλίου λοιπόν, το οποίο βασιζόμενο σε ανεξάρτητες αναλύσεις θα μπορούσε να προχωρήσει σε ανάλυση της συνοχής των διαφόρων προϋπολογισμών στο πλαίσιο των κανόνων σταθερότητας και ανάπτυξης και να αναζητήσει για χώρες οι οποίες πληρούν τους όρους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ε, περιθώρια για να συμβάλλουν στην ανάπτυξη μακροοικονομικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν χώρε οι οποίες έχουν μεγάλο πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών ε, και θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη σταθεροποίηση το, της Ευρωζώνης. Αυτός ο συντονισμός θα ήταν ένα κεντρικό στοίχημα. Θα πρέπει να προβληθεί ως ε, αναζήτηση, σε μια συζήτηση με ένα ανεξάρτητο, όπως είπα, συμβούλιο, το οποίο σε μια πρώτη φάση θα έπρεπε, χωρίς να τροποποιηθούν οι συνθήκες, σημειώνω, να υποβάλει συστάσεις που θα συζητούσαν συνέχεια τα θεσμικά όργανα, όπως υπάρχουν το Κοινοβούλιο, το ε, Eurogroup κτλ. ώστε να ανοίξει και να επηρεαστεί και η σχετική συζήτηση στα εθνικά κοινοβούλια που θα οδηγούσαν προς τον εθνικό συντονισμό. Στον, στον ε, συντονισμό καλύτερα των εθνικών προπολογισμών. Αλλά, αλλά αυτό παραμένει αυτή τη στιγμή ως αδύναμπτο εγχείρημα μέσω πρόθεσμα. Ήταν τόσο δύσκολο ο συντονισμό των νομισματικών πολιτικών πριν την Ευρωζώνη που χρειάστηκε να συσταθεί η Ευρωζώνη για να εξασφαλίσει ο συντονισμό, ε, ο συντονισμό των εθνικών προπολογισμών θα σήμαινε υπέρβαση των εθνικών προπολογισμών που θα πρέπει να συντονιστούν βέβαια στο μέγιστο δυνατό βαθμό, αλλά πάλι με τα όρια. Οπότε θα χρειαζόταν ένα αντικυκλικό δημοσιονομικό εργαλείο μέσα σε αυτή την Ευρωζώνη. Αυτό το δημοσιονομικό εργαλείο που υπενθύμησε και ο κύριο Κνότ, ε, θα πρέπει να ε, ανταποκρίνεται σε μια σειρά από κριτήρια αντιμετώπιση δυσχεριών και προκλήσεων και του ηθικού κινδύνου και της ενθάρρυνσης προσφέλτησης πρακτικές σε εθνικό επίπεδο και ως προς την συμβατότητά του σε σχέση με τα νομοθετήματα, τα θεμελιώδη των κρατών μελών και όλα αυτά βεβαίως δεν μπορούν και να αποκρύψουν την αναγκαιότητα και τη δυνατότητα προσδιορισμού ενός τέτοιου εργαλείου εφόσον το επιτρέπουν, ε, επιτρέπουν τον προσδιορισμό του τα σχετικά ε, στοιχεία. Ένα τέτοιο λοιπόν εργαλείο που έχουν κοινοτοποιήσει άλλε ομοσπονδίε συμβατό με τι ιδιαιτερότητε εθνικέ που αναφέρθηκαν και νωρίτερα και που συζητούνται αυτή τη στιγμή, καλύπτεται μαζί παράλληλα με μια ευρωπαϊκή ασφάλιση ανεργία που θα μπορούσε να χτιστεί μέσα στην Ευρωζώνη και θα αποτελούσε ένα δημοσιονομικό αντικυκλικό εργαλείο τη Ευρωζώνης. Πολλέ λύσει προτείνονται για αυτή την ευρωπαϊκή ασφάλιση ανεργία. Ε, πάλι με απόλυτο ρεαλισμό και πραγματισμό σε σχέση με διάφορες άλλες νομισματικές ε, ομοσπονδίες. Θα προβάλλω το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών ως νομισματικής ομοσπονδίας που επιτρέπει το συνδυασμό ενός εργαλείου ομοιογενειοποίησης ε, γιατί είναι πολύ μεγάλος αυτός, πολύ έντονος αυτός ο χαρακτήρας 0,3 με 0,6 είναι το το αναπλήρωσης που υπάρχει σε ομοσπονδιακό επίπεδο σε σχέση με τις πολιτείες, άρα είναι κάτι το ζητούμενο αντίστοιχα και για την Ευρωζώνη, Αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε έναν ευρωπαϊκό, έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ομοσπονδιακό που θα επέτρεπε την αποζημίωση των μακροπρόθεσμα ανέργων σε υψηλό επίπεδο, ιδιαίτερα, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τη κάθε χώρα, χρηματοδοτούμενο από το ευρωπαϊκό επίπεδο στο ευρωπαϊκό επίπεδο, σε περίπτωση κρίσεω για κάποια συγκεκριμένη χώρα που θα πλήττεται από μια κρίση, με, αντίστοιχο, αντίστοιχη στάθμιση τη αύξηση του ποσοστού ενεργεία. Χωρί να μπαίνω στι ιδιαιτερότητε τεχνικέ αυτή τη ε, ιδέα μια ασφάλισης ενέργεια και τρόπου θέσπισής γιατί υπάρχουν πολλέ λύσει που προτείνονται Πιστεύω ότι για να προχωρήσουμε σε αυτή τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού προϋπολογισμού πρέπει να μας απασχολήσει το ζήτημα ενός συγκεκριμένου εργαλείου συμβατού με τις ιδιαιτερότητες της Ευρωζώνης και τις ετερογένειες που μπορεί να χαρακτηρίσει και αυτό θα ήταν το καλύτερο μέσο να μια ασφάλιση ενεργείας δηλαδή. Που θα ακολουθεί τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αυτή η ασφάλιση ενεργείας θα επέτρεπε σταθεροποίηση των κινδύνων σε επίπεδο Ευρωζώνης αν όμως είναι μακροοικονομικός ο κίνδυνος, ε, η δυνατότητα για ανάληψη χρέους σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να είναι και δυνατή χάρη σε ομόλογα που θα επέτρεπαν αντικυκλικά τη διαχείριση του μακροοικονομικού κινδύνου. Και θα σταματήσω εδώ για να μην ξεπεράσω το χρόνο μου, υπενθυμίζοντας τις τρεις σημαντικές διαστάσεις, να ληφθεί υπόψη δηλαδή η διάσταση της σταθεροποίησης της ζήτησης και εντοπισμό, χαρακτηρισμό αυτής ως αιτία της μη τήρησης μετά την κρίση των κανόνων που είχαν προβλεφθεί για το συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών ε, των κρατών της Ένωσης. Δεύτερον, πραγματισμό και ρεαλιστική σύγκριση με άλλες νομισματικές ενώσεις ή ομοσπονδίες. Και τρίτον, πρόοδο ε, συντονισμένη προς ένα κοινό εργαλείο ασφάλισης ανεργίας στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Ραγκού για τις εξηγήσεις σας, για το φως που ρίξατε στην υπόθεση και τώρα παρακαλώ τους δύο συγκητές μας που θα απαντήσουν, θα αντιδράσουν στις τρεις ομιλίες, θα σχολιάσουν και θα θέσουν και ερωτήσεις. Ο κύριος Μπόγκε. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ κύριε Εκρό για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Αναφερθήκατε και ξεκαθάρισατε δύο συγκεκριμένα πράγματα πολύ σημαντικά. Πρέπει να ολοκληρωθεί η οικονομική και νοσηματική έρωση παρά την κρίση και παρά τις ε, μεγάλες προκλήσεις με των οποίων βρισκόμεθα. Ε, και αυτό το λέω σημειώνοντα ότι αν δεν μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την αποκατάσταση αλληλεγγύη και τη συνεργασία στα κράτη-μέλη, δεν θα το καταφέρουμε αυτό ποτέ. Δεύτερον, είπατε χωρίς στήριση των ε, κοινών κανόνων δεν μπορεί να προκύψει ε, εμπιστοσύνη. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο νομίζω όταν μιλούμε για τέτοιου είδους εργαλεία που μπορούν να μας βοηθήσουν να διαφυλάξουμε τη σταθερότητα του ευρώ σε συνθήκες πλαισίου και ταυτόχρονα σε παγκόσμιο επίπεδο να του επιτρέψουμε να έχει πιθανότητες ε, επιβίωσης. Αλλά βέβαια τότε Πρέπει να ξεφύγουμε ίσως από την ιδέα των κυριαρχών κρατών και θα συμπληρώσω ότι και στο ευρώ σε ορισμένα σημεία της δημοσιονομικής πολιτικής για καταπιστεύματα ή για έκτακτη ανάγκη, μέτρα έκτακτης ανάγκη τα οποία βεβαίως και θα πω ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε και θα τα χαιρετήσω. Ε, βρισκόμαστε στο outsourcing και όχι στην κοινοτική μέθοδο και πρέπει εδώ να καταστήσουμε σαφές ότι οι τέσσερις βασικές ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς ε, προβλέπουν και μαζί με, όλοι, με τις τέσσερις ελευθερίες έχουμε ως κανόνα το ευρώ και όλα τα υπόλοιπα είναι εξαίρεση. Οπωσδήποτε είναι έξω το ευρώ, πρέπει να τίνει προς το ευρώ και αυτό ακριβώς είναι και ο πυρήνας και γι' αυτό δεν θα πρέπει να έχουμε αυτό το outsourcing την όλο και πιο έντονη διακυβερνητική ε, διαχείριση που βλέπουμε και που επιδεινώνει διαρκώς την κατάσταση. Και επίσης, Υπάρχει μια εξέλιξη όπως αναφέρθηκε που θα οδηγούσε στον περιορισμό των κινδύνων για τις τράπεζες και αντίστοιχα και για τον φορολογούμενο. Ερωτώ λοιπόν, αυτοί, αυτές οι λύσεις έχουν προχωρήσει αρκετά και επίσης η δημοσιονομική ικανότητα σε σχέση με τα υφιστάμενα εργαλεία. Το μηχανισμό σταθερότητας, το αδερφωτικά ταμεία, το ταμείο συνοχής, το οποίο έχει συγκεκριμένο στόχο ε, όταν ιδρύθηκε η πρωτοβουλία για την ε, πασχόληση των νέων. Με αυτά τα εργαλεία λοιπόν βλέπετε να εξασφαλίζονται οι στόχοι. Και επίσης αμέσως μετά από αυτά προκύπτει και το ερώτημα πώς αυτή η δημοσιονομική ικανότητα αναπτύσσεται και αν αναπτύσσεται μόνο για τα ε, κράτη της Ευρωζώνης και για τα κράτη εκτός Ευρωζώνης όπως είχε αναφερθεί από το 2011 και επίσης αν δεδομένης οικονομικής και πολιτικής κατάστασης μέσα στην οποία κινείται η Ευρωζώνη μπορεί να υπάρξει ένας σχεδιασμός σταδιακός που να προχωρήσει και ταυτόχρονα με απόδειξη του κάθε σταδίου ότι έχει τηρηθεί, για το κάθε στάδιο ότι έχει τηρηθεί το σύνολο των προϋποθέσεων προκειμένου να προχωρήσουμε στο επόμενο, έτσι ώστε να ανακτηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη και έτσι να ενισχυθεί η προοπτική για μια καλύτερη δημοσιονομική ικανότητα στο τέλος της Ευρωζώνη. Ευχαριστώ. Merci, Σας ευχαριστώ κύριε Μπέγκε. Κυρία Μπερές, ευχαριστώ. Τηλεγραφικά θα θέσω τις ερωτήσεις μου. Ε, κύριε Μπενουά Κερέ, μιλήσατε για σταδιακό χαρακτήρα και ε, αιρεσιμότητα. Έχουμε όμως το χρόνο για κάτι τέτοιο. Αφήστε την προσφυγική κρίση, αφήστε τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ας επικεντρωθούμε μόνο στην κατάσταση όπου η νομισματική μας πολιτική έχει φτάσει στα όρια της σχεδόν. Ναι. Και το θέμα των επιτοκίων κάνει τον αντίκτυπο της νομισματικής πολιτικής στην οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης περιορισμένο. Περιορίζει αυτόν τον αντίκτυπο. Αλλά διαπιστώνουμε ότι οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ε, διευρύνονται και οξύνονται. Μας είπατε ότι οι πολιτικοί θα πρέπει να λάβουν τις αποφάσεις, αλλά παρόλα αυτά δεχτήκατε να λάβετε μέρος στην ακρόαση. Επιμείνατε στο θεσμικό σκέλος, στις θεσμικές πτυχές ενός μηχανισμού που θα πρέπει να συνοδεύει την ε, δημιουργία προϋπολογισμού της Ευρωζώνης. Εδώ στο έγγραφο εργασία μας ε, υπάρχουν πολλές προτάσεις. Μία από αυτές προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνει το κοινοβούλιο που θα αξιολογεί τον προϋπολογισμό της Ευρωζώνης αν υπάρχει τέτοιο ειδικό προπολογισμό Ευρωζώνης. Θεωρείτε ότι είναι σκόπιμο κάτι τέτοιο. Είναι μια καλή λύση. Κύριε Κνότ, έχω δύο ερωτήσεις για σας. Ερώτηση πρώτη. Αναφερθήκατε εν παρόδο στον ε, μηχανισμό ε, εποπτείας των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Θεωρείτε ότι αξιοποιούμε δεόντως αυτό το μηχανισμό και την ανάλυση του ή μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε περισσότερο. Δεύτερη ερώτηση. Αφορά την τέταρτη σας παρατήρηση. Είπατε ότι με, την, με τον ιδιωτικό επιμερισμό των κινδύνων μπορούμε να καταλήξουμε σε εξίσου ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Και συγκρίνεται την κατάσταση της Ευρωζώνης με την κατάσταση της Ηνωμένες Πολιτείες ε, ή στη Γερμανία. Στι δύο όμω αυτέ τι περιπτώσει, είπα και η Γερμανία, και είναι κάπω παράδοξο που χρησιμοποιείτε αυτά τα δύο παραδείγματα, γιατί και στα δύο παραδείγματα ο μηχανισμό προστασία, το backstop, και το θέμα του προπολογισμού που μπορεί να στηρίξει και τον ιδιωτικό κίνδυνο αν, αν παρουσιαστεί υπάρχει υπάρχει αυτή η δυνατότητα και όλη η συζήτηση που γίνεται γύρω από την Ένωση Κεφαλαγορών Αφήνοντα να εννοηθεί ότι αν αναπτύξουμε την Ένωση Κεφαλαγορών θα έχουμε καλύτερη πρόσβαση των οικονομικών τελεστών στις χρηματοπιστωτικές αγορέ, οπότε θα αντισταθμίσουμε τη δυσκολία εφαρμογής μιας δημοσιονομικής πολιτικής. Αν αναφερόμαστε όμως ε, στην Ένωση Κεφαλαγορών, μία προϋπόθεση για να λειτουργήσει η Ένωση Κεφαλαγορών είναι να ολοκληρώσουμε πρώτα την Τραπεζική Ένωση και επανερχόμαστε στο θέμα του μηχανισμού προστασίας που χρειάζεται και για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και για την αξιόπιστη θέσπιση της Ένωσης Κεφαλαγορών. Είναι σαν να έχουμε ένα γάτο που προσπαθεί να και προσπαθεί να δακώσει την ωρά του. Τώρα, η χρήση της νομισματικής πολιτικής σε μια περίοδο μεγάλης έντασης είναι κάτι στο οποίο και εμείς έχουμε σκοντάψει. Πώς μπορούμε επίσης να καταστήσουμε αξιόπιστη τη διαδικασία σύγκλησης θα βάλω τελεία κύριε Πρόεδρε, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που συζητήθηκε εκτενώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την ιδέα ενός κώδικα σύγκλησης κατά το πνεύμα των κριτηρίων του Μάστριχτ ώστε να έχουμε έναν ορισμό μέσα σε μια πενταετία δύο-τριών στόχων που οφείλουν να υλοποιούν τα κρατημέλη για να προσδιορίσουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με μεγαλύτερο ownership εκ μέρου από ότι σήμερα. Ευχαριστούμε κύριε Μπερέ. Ο λόγο στου εμπειρογνώμονέ μας, τους καλεσμένους μας και τους θερμοπαρακαλώ αν γίνεται να περιοριστούν σε ένα δίλεπτο. Κύριος Κερέ, δύο λεπτό καθένας εννοείται. Συγγνώμη, αλλά έχω πρόβλημα με τη φωνή μου. Θα ξεκινήσω με τις απαντήσεις προς την κυρία Μπερές. Πόσο επιτακτική είναι ανάγκη, πόσο επίγουσα και η σταδιακή και η πόρου σύγκληση. Φυσικά είναι και κατεπήγον το θέμα. Επιτακτική ανάγκη. Δεν θα έλεγα ότι έφτασε στα όρια της η ένωση. Δεν είναι αυτό το αντικείμενο της σημερινής συζήτησης, αλλά συμφωνώ. Όσο οι υπόλοιπε πολιτικές και οι δημοσιονομικοί μπορούν να συμβάλλουν στην ανάκαμψη, ε, τόσο το καλύτερο για μας. Θα ελαφρύνει το βάρος ε, της δημοσιονομικής πολιτικής που σήμερα είναι τεράστιο. Υπάρχει λοιπόν επίγουσα ανάγκη. Και χρειάζεται τουλάχιστον αυτή τη διαδικασία σύγκληση για τον απλούστατο λόγο να αποφύγουμε η δημοσιονομική, αυτή η κοινή δημοσιονομική ικανότητα να, να μετατραπεί σε μονόδρομε μεταφορέ. Γιατί αυτό δεν υπακούεται στο πνεύμα ούτε στο γράμμα τη συνθήκη, ούτε στο σύμφωνο ίδρυση τη ΟΝΕ δεν ε, έγινε η ΟΝΕ για μονομερείς μόνο, μονόδρομες ε, ε, μεταφορές προς τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν δυνατότητες μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, ταμείων συνοχής και το καθεξής, αλλά δεν είναι το αντικείμενο αυτή τη συζήτηση. Σε ό,τι αφορά το θέμα της δημοκρατικής ευθύνης, δεν θα διακινδύνευα μια συζήτηση για το ποιο θα πρέπει να είναι ο σχετικό ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ΕΚΤ φυσικά είναι στο πλευρό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πάντα, λόγω της φύσης της, αλλά θα εξαρτηθεί και από τον τρόπο με τον οποίο θα συγκροτηθεί αυτή η δημοσιονομική ικανότητα. Και για να γίνει αποδεκτή πολιτικά, θα πρέπει να προβλέψει κάποιο ρόλο και για τα εθνικά κοινοβούλια. Δεν είναι εύκολη ερώτηση, γι' αυτό και δεν υπάρχει εύκολη απάντηση. Για τις ερωτήσεις του κ. Μπέγκε και φαίνεται ότι θα ξεπεράσω το δίλεπτο, κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Μπέγκε μίλησε κυρίως για την κοινοτική μέθοδο. Πολύ σημαντική στη συζήτηση η διαπίστωση και η επιβεβαίωση ότι κάθε μηχανισμό που θα δημιουργηθεί μετά τη συζήτηση, ω απόρρια τη συζήτηση, θα πρέπει να ενταχθεί στην κοινοτική μέθοδο. Και αν μπορέσουμε να επαναντάξουμε κάποιου μηχανισμού που δεν είχαν υπαχθεί αρχικά στην κοινοτική, καλό θα ήταν. Για παράδειγμα, το μηχανισμό σταθερότητα. Αυτό είναι πραγματικά ευκταίο και επιθυμητό. Και θα επιτρέψει και στο Κοινοβούλιο να αναλάβει το ρόλο του. Σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ κινδύνου δημόσιου χρέους και τραπεζικού κινδύνου, θα πρέπει να γίνει αποσύνδεση των δύο κινδύνων. Αυτό θα γίνει σταδιακά και μέσω πρόθεσμα. Για παράδειγμα, υπάρχει μια οχταετία. οχταετή είναι για το Ταμείο Εξυγείας των Τραπεζών. Οπότε έχουμε μια σταδιακή, ένα σταδιακό χαρακτήρα και επίσης να περιορίσουμε την έξεση των τραπεζών στο δημόσιο χρέος. Και αυτό θα γίνει σταδιακά και στο μέτρο του δυνατού θα πρέπει να γίνει με τρόπο συνεκτικό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Κάτι που προϋποθέτει φυσικά εκτενέστατες συζητήσεις. Ευχαριστούμε κύριε Κέρε, ο πρόεδρος Κνότ. Yeah, thank you σας ευχαριστώ για τις τόσο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Θα είναι πραγματική πρόκληση να τις απαντήσω όλες σε δύο λεπτά. Αλλά να ξεκινήσω από τις ερωτήσεις της κυρίας Μπερές. Οι μακροοικονομικές ανισορροπίες και σχετική διαδικασία κατά πόσον την αξιοποιήσαμε παρκώ. Να σα δώσω μερικού αριθμού. Η διαδικασία είναι σχετικά πρόσφατη. Όμω ήδη έγινε μια αξιολόγηση τη πρώτη χρονιά εφαρμογή τη. Πολλέ είναι οι συστάσει που προέκυψαν μετά την πρώτη χρονιά, αλλά από αυτέ μόνο 5% έγιναν σεβαστέ από τα κράτη-μέλη. 50% των συστάσεων ε, γνώριζαν κάποια συνέχιση και κάποια εφαρμογή από τα κατημέλη και το υπόλοιπο 45% όλων των συστάσεων δεν λήψαν καθόλου υπόψη. Εάν δείτε αυτού του αριθμού, αυτά τα ποσοστά, τουλάχιστον από τη δική μου τη σκοπιά, νομίζω ότι δεν αξιοποιούμε πλήρω το δυναμικό τη διαδικασία. Και αυτό πραγματικά αποκαλύπτει ένα πρόβλημα για τον τρόπο που η Ευρώπη αντιμετωπίζει τους κανόνες που η ίδια σχεδιάζει για τον εαυτό τη. Ο ίδιος ο σχεδιασμός των κανόνων είναι ένα θέμα διαφορετικό από το πώς υλοποιούνται και το πώς εφαρμόζονται. Και οι κανόνες υπάρχουν με ένα επιχάρτου ε, στο, στη θεωρία, αλλά μετά στην πράξη δεν ε, τηρούνται. Οπότε ε, είναι δύσκολο να δημιουργηθεί ένα, το απαραίτητο κλίμα εμπιστοσύνη. Την εμπιστοσύνη που επεκαλέστηκαν και οι συναδελφοί σα για να υπάρξει μια διαδρομή, μια πορεία σταδιακή ανοικοδόμηση, ανάκτηση τη εμπιστοσύνη. Πώ λοιπόν να περάσουμε σε μεταρρύθμιση τη κατανομή του κινδύνου, διότι ο βαθμό κατανομή του κινδύνου αυτή τη στιγμή ε, στην Οικονομική Νοσματική Ένωση δεν επαρκεί. Είναι σαφέ νομίζω αυτό. Δεν συμφωνήσαμε αυτή την Οικονομική και Νομισματική Ένωση το 1999. Ε, δεν ήταν απλώς νομισματική. Ε, μάλλον ξεκίνησε απλώς ως νομισματική, αλλά άλλες βλέψεις είχαμε. Δεν θα πρέπει λοιπόν κάτι να γίνει ε, πέρα από αυτή τη βαθμία προσέγγιση, διότι Ούτε πιο γρήγορα από ό,τι επιτρέπει η διαδικασία μπορούμε να πάμε, γιατί έτσι θα δημιουργηθεί απαραίτητη εμπιστοσύνη για την κατανομή των κινδύνων, για την Τραπεζική Ένωση και ε, για την ε, σύνδεση των τραπεζών με τα κρατικά χρέη. Ναι, εδώ υπάρχει το θέμα της εγγύησης των καταθέσεων, του μηχανισμού προστασίας backstop, αλλά και του μηδενικού κινδύνου ή της προτιμησιακής μεταχείρισης κινδύνου στους ισολογισμούς για τα κράτη-μέλη και τα κρατικά τους χρέη, τα κάτι που δεν μπορούν πλέον να δώσουν δικό τους νόμισμα, να κόψουν δικό τους νόμισμα. Οπότε θα πρέπει να το δούμε και από τις δύο όψεις. Όταν ε, η τριγμή της χρηματοοικονομικής αγοράς ε, ε, ηρέμησαν στην αρχή της φετινής χρονιάς, είδαμε τι γίνεται μεταξύ των spread των τραπεζών και τον συσχετισμό τους με το κρατικό χρέος. Και πάλι ήρθαν πιο κοντά. Άρα δεν έσπασε ο δεσμός αρκετά, δεν χτυπήθηκε όπως έπρεπε. Εκεί πρέπει να δώσουμε ένταση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ραγκό. Ναι, ευχαριστώ και εγώ πολύ γρήγορα μερικές παρατηρήσεις. Συμπληρωματικά. Και καταρχά για τα όρια της νομισματικής πολιτικής υπάρχει ένα σημείο το οποίο πρέπει νομίζω να σημειώσουμε η νομισματική πολιτική είναι ετερογενή στην Ευρωζώνη σήμερα, όπως και η ικανότητα των τραπεζών να βρουν λύσεις ε, σε περίπτωση που μετακομίζουμε στην Ευρωζώνη ε, επιχειρήσεις για τις οποίες δεν μπορούν να βρουν λύσεις οι τράπεζες. Άρα λοιπόν θα υπάρχει και ένας σταθεροποιητικός παράγων και μπορούν έτσι να βρουν μια ομοιογένεια ε, μέσα στη ζώνη ευρώ χάρη στη σταθεροποίηση αυτή. Ένα δεύτερο σημείο, ο προϋπολογισμός ο απαραίτητος για τη σταθεροποίηση. Ο, δημοσ... ο προϋπολογισμός ομοσπονδιακός ε, δεν ε, πρέπει να είναι χαμηλότερος από το 6% γιατί είναι πολλές από τις ε, λειτουργίες των προϋπολογισμών αυτών των ομοσπονδιακών σημαντικές τόσο και κυρίαρχες θα λέγαμε που δεν μπορούν να καλυφθούν από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Ένας μικρός λοιπόν προϋπολογισμός ομοσπονδιακός, 2-3% επί του ΑΕΠ της Ευρωζώνης, μπορεί να συμβάλλει σταθεροποιητικά αφού όλες αυτές οι κυρίαρχες εξουσίες μακροπρόθεσμα θα παραμένουν στα χέρια των κρατών μελών. Η επιχειρηματολογία δηλαδή της ε, ε, σταδιακής εισαγωγής ενός ε, ευρωπαϊκού προϋπολογισμού δεν θα πρέπει, ενός προϋπολογισμού της Ευρωζώνης δεν θα πρέπει να ε, υποτιμά και τη σημασία της, παρεμβάσης, ε, της δυνατότητας παρέμβασης ενός μικρότερου ομοσπονδιακού προϋπολογισμού σταθεροποιητικά ε, ως δε μέσον εξασφάλιση μιας σύγκλησης στην αγορά εργασίας αυτή η ασφάλιση ανεργίας μπορεί να ε, ε, απαντηθεί ως εξή. Υπάρχει μεγάλη ετερογένεια και πριν αλλά και μετά την κρίση στις αγορές εργασίας στην Ευρωζώνη. Άρα πρέπει να συγκλίνουν αυτές. Κάποιοι μπορεί λοιπόν να χάσουν ανταγωνιστικότητά τους, να χρειάζονται μεταρρυθμίσεις διαστρωτικές. Αυτό το μέτρο λοιπόν σταθεροποίησης είναι συμπληρωματικό της σύγκλησης στην αγορά εργασίας της Ευρώπης. Άρα ένας κώδικας σύγκλησης, πενταετής, που θα οδηγήσει σταδιακά στη σύγκληση προς τα άνω, όχι υπό, όχι υποπληθωριστικά, όχι οδηγώντας δηλαδή σε ελλείμματα περισσότερο, μη, υπο, μη ε, αποπληθωριστικά σύγκληση πρέπει να γίνει και βέβαια πολύ σταδιακά, ανάλογα και με τη ζήτηση και όλα αυτά, μια προστάνω λοιπόν σύγκληση, μια ε, ασφάλιση ενέργειας που θα εξασφαλίσει μια σύγκληση και των αγορών εργασία και, και, θα αυτό σε συνεργασία με ένα μικρό προπολογισμό, νομίζω ότι θα οδηγήσει, θα οπίσει τη ζώνη σε ευρώ. Ευχαριστώ ο κύριος Γκουαλτιέρη, ήρθε ο πρόεδρος. Εν τω μεταξύ είχαμε συμφωνήσει ώστε να λάμβανε εκείνο τα ενία της συνεδρίασης επιστρέφοντας, Ρομπέρτο. Για να δούμε και τους κοιόδης τώρα. Παρακαλώ. Ο κύριος Μούρεσαν. Ευχαριστώ τους συμπροέδρους και τους καλεσμένους μας για τις πολύ χρήσιμες ε, πληροφορίες που μας έδωσαν. Το θέμα είναι γιατί χρειαζόμαστε τη δημοσιονομική ικανότητα και δεδομένων των οικονομικών περιορισμών που έχουμε και της δυσπραγίας, ε, τι μπορούμε να κάνουμε. Χρειαζόμαστε ένα τρόπο να απορροφούμε τα σοκ, τους κρατασμούς συμπληρώνοντας την Τραπεζική Ένωση ή να δώσουμε κίνητρα για διαστροτικές μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα. Και απευθύνω κυρίως την ερώτηση στους δύο εκπροσώπους ε, των κεντρικών τραπεζών, γιατί οι κεντρικοί τραπεζίτες, οι διοικητές κεντρικών τραπεζών μίλησαν για την ανάγκη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Τι μεταρρυθμίσεις θεωρείτε ότι είναι απαραίτητες για να συμπληρώσουν τα μέτρα της νομισματικής πολιτικής που έχει ε, εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και χρειάζονται και κάποια χρηματοοικονομικά κίνητρα. Γιατί θέλουμε φυσικά τη δημοσιονομική ικανότητα τη Ευρωζώνη να τη συνδέσουμε με ρεσιμότητα, με ισχυρέ προποθέσει. Αλλά οι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει δεν κοστίζουν χρήματα και επηρεάζουν αρνητικά την δημοσιονομική θέση των κρατών μελών ε, ή όχι. Και κατά τη γνώμη μα, τι, τι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει χρήζουν και δημοσιονομικών κινήτρων σε ό,τι αφορά τι χώρε εκτό Ευρωζώνη, πώ μπορούν και αυτέ να ενταχθούν στην δημοσιονομική ικανότητα και πώ μπορούν να αξιοποιήσουν τα ωφέλη πριν να ενταχθούν στην ΟΝΕ. Ποια θα ήταν τα ωφέλη των χώρων εκτό Ευρωζώνη από τη συμμετοχή του στη δημοσιονομική ικανότητα και ποια τα μειονεκτήματα ή τι διαβεβαιώσει θα μπορούσαμε να δώσουμε στι χώρε εκτό Ευρωζώνη μετά τι παραχωρήσει που κάνουμε και στην Μεγάλη Βρετανία ε, και τις χώρες εκτός Ευρωζώνης που δεν θέλουν να ενταχθούν στο ευρώ, τι ε, διαβεβαιώσεις ε, θα δώσουμε ότι η ενίσχυση της δημοσιονομικής ικανότητας δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες σε χώρες εκτός Ευρωζώνης. Επίσης, είπατε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς που έχουμε ώστε τα κράτη-μέλη που συμμορφώνονται με το δημοσιονομικό σύμφωνο να λαμβάνουν κάποια ανταλλάγματα. Ποια είναι τα μέτρα που προτείνετε για να ενισχύσουμε αυτή τη διαδικασία. Η κυρία Πύρκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για τα πολλά, πολύ ενδιαφέροντα σχόλια και τις απόψεις που παρουσιάσατε. Όπως είπαν οι συνεισηγητές μας, η δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης είναι κάτι που έχει ήδη συζητηθεί στο παρελθόν. Κατά τη γνώμη σας, είναι ρεαλιστικό τα κράτη-μέλη να ταχθούν υπέρ ενός τέτοιου μηχανισμού. Επίσης, πού βρίσκονται τα προβλήματα των κρατών μελών και τι αντίκτυπο θα έχει ένας τέτοιος μηχανισμός δημοσιονομικής ικανότητας στην κυριαρχία των κρατών μελών. Επίσης, ε, ποιο θα ήταν το κατάλληλο χρονικό σημείο για την δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ κύριο Σαρτουί. Ο κύριος Κερέ μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκανε το καθήκον της και μάλιστα μερικές φορές ξεπέρασε και την ειδική της αποστολή και βοήθησε εκεί που δεν υπήρχε οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη. Προσπάθησε να καλύψει αυτό το κενό. Ας μην κρυβόμαστε λοιπόν πίσω από το δάχτυλό μας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο προϋπολογισμός είναι απλώς η έκφραση μιας ικανότητας και μιας πολιτικής βούλησης. Δεν μπορούμε να φανταστούμε έναν προπολογισμό χωρίς πολιτικό όραμα που να τον στηρίζει. Και θα πρέπει να αντλήσουμε τα διδάγματα από το γεγονό ότι ε, έγινε ένας επιμερισμός της ε, ε, δημοσιονομικής, κυριαρχία. οικονομικής κυριαρχίας και δεν υπάρχει πώληση μίξ, δεν υπάρχει μείγμα πολιτικό γιατί δεν υπάρχει τέτοια δημοσιονομική ικανότητα. Υπάρχει ένας τρόπος ε, επιμερισμού του, της υπερχρέωσης των χωρών της Ευρωζώνης ώστε να αντιμετωπιστούν τα ασύμετρα σοκ, οι ασύμετροι καταδασμοί. Επίσης, τι αρμοδιότητες θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε από τα κράτη-μέλη στην Ευρωζώνη. Ο κύριος Αρμό μίλησε για την ασφάλιση ανεργίας. Τι κοστίζει τα κράτη-μέλη η συμμετοχή σε μια τέτοια πολιτική. Αν αυτό μεταφερθεί στην Ευρωζώνη, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν με αντίστοιχο ποσό από αυτό που θα έπρεπε να πλήρωναν από μόνο τους αν δεν υπήρχε αυτή η αρμοδιότητα. Τι άλλες αρμοδιότητες θα μπορούσαν να μεταφερθούν στην Ευρωζώνη ώστε να γίνει πιο ισχυρός ο προϋπολογισμός ελαφρύνοντας κάπως τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα λάβει χώρα και η σύγκληση και η Ευρωζώνη θα γίνει η αυτή η άριστη νομισματική περιοχή που επιθυμούμε όλοι και από την οποία ακόμη πόρο απέχουμε. Ο Φάμπιο Ντεμάζη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, αναφέρθηκε σε διάφορες ε, εκθέσεις και μια πλημμύρα από εμπειρογνωμοσύνες για να προσπαθήσω και εγώ να αναφερθώ σε αυτά. Αναφερθήκατε σε ανεπαρκή δράση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Θέλω να πω ότι η Ισπανία και η Ιρλανδία είχαν το χαμηλότερο ποσοστό προσαρμογής επί του ΑΕΠ και δεν νομίζω ότι αυτό εξηγεί ότι υπάρχουν ιδιωτικοί μηχανισμοί από ρόφηση ε, κινδύνων, γιατί έχουμε δει να κυκλοφορούν διάφορα χαρτοφυλάκια. Αναφερθήκατε στον Ρόμπερτ Σίλερ Φερρυπίν που είχε κερδίσει και το βραβείο Νόμπελ, που είχε τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ, αναφερόμενος στις ε, αδυναμίες των κεφαλαϊκών αγορών για απορρόφηση των ε, σοκ αυτών των διδονισμών. Αλλά για να δω αν ο κύριος Ραμπό μπορεί να μου απαντήσει δύο ερωτήσεις. Συμφωνώ ότι η δημοσιονομική ικανότητα είναι κάτι το πολύ δύσκολο, δεν θα εξασφαλίσει δηλαδή συνένεση εύκολα. Υπάρχουν ζητήματα διαφιλονικούμενα, δεν είναι σταθερή πηγή χρηματοδότησης, η φορολογία. Τι θα βλέπατε λοιπόν εσείς, γιατί βλέπουμε ότι η δημοσιονομική πολιτική εξουδετερώνεται από την υπερβολική δημοσιονομική πειθαρχία, δεν μπαίνει το χρήμα στην πραγματική οικονομία και άρα αυτό εξωτερώνει ε, τα ωφέλη της χρήσης ενός αρνίου συστήματος. Και επιπλέον θα ήθελα να πω ότι θα μπορούσε να πέσει και το επίπεδο φορολόγησης για τον πολίτη, εάν βοηθούσαν χώρες όπως οι κάτω χώρες και αν συνέβαλαν και στη δουλειά μας που κάνουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ένα πιο δίκαιο σύστημα φορολογικό για τις επιχειρήσεις Φερρυπίν. Ε, επίσης ο κύριος Στίγλιτ σε εβδομάδε εβδομάδες επισκεφθεί τις Βρυξέλλε για να μιλήσει για του χρυσού κανόνα των επενδύσεων. Δημόσιε επενδύσει, δηλαδή θα πρέπει να αποκλείονται από του κανόνε περί ε, χρέους των κρατών γιατί αποτελούν επένδυση, δηλαδή πλούτο για τις επόμενες γενιές. Το ίδιο συμβαίνει και με τον αντίστοιχο νόμο για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της Γερμανίας. στα και τέτοια. Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά. Ριάντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να είμαστε σύντομοι γιατί έχει αναφερθεί πολλές φορές. Είναι ε, λιγότερο από 1% ο προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ΑΕΠ όλων των χωρών της ε, Ευρώπης. Η όξυνση των ισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και η έλλειψη αλληλεγγύης καθώς και μηχανισμών επίδειξης αυτής δείχνουν ότι δεν μπορούμε να επαφήσουμε τις ελπίδες μας στο δημοσιονομικό πλαίσιο και τις δημοσιονομικές δυνατότητες όπως διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει καχυποψία, όπως βλέπουμε, μεταξύ των κρατών και των εταίρων τους ήδη. Ε, τα πιο αδύναμα κράτη-μέλη τελικά πληρώνουν το τίμημα της αλληλεγγύης με τη λιτότητα και η αστάθεια συνεχίζεται στην Ιρλανδία. Το είδαμε πολύ πιο έντονα από ό,τι άλλε χώρε, όπου κάθε άντρα, γυναίκες και, γυναίκα και παιδί θα πληρώνουν χιλιάδε επί χιλιάδων ευρώ τα επόμενα 50 χρόνια για να ξεπληρώσουν όσα έγιναν. Ε, δεν μπορούμε λοιπόν να ανακτήσουμε εύκολα την εμπιστοσύνη στα κράτη-μέλη. Πιστεύετε λοιπόν ότι μπορούμε να έχουμε τέτοιε θεωρητικέ και αφηρημένε δομέ σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση για να ζήσουν οι άνθρωποι με ελπίδα. Έχω πολλέ αμφιβολίε και σοβαρέ. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε λοιπόν μια τέτοια τραπεζική κρίση στο μέλλον ε, μια δημοσιονομική και τραπεζική κρίση. Και τι μπορεί να γίνει άμεσα στα πλαίσια της Τραπεζικής Ένωσης που εσείς περιγράψατε. Ευχαριστούμε ε, ο κ. Μαραγκάλη. Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε θα μιλήσω ισπανικά. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Αρτουή. Επίσης ενστενίζομαι αυτά που είπε ο κύριο Δεμάζη για την εξέλιξη του ισπανικού χρέους. Δεν θα επιμείνουμε, απλώς διαπιστώνουμε αυτή την κατάσταση. Τέσσερα συγκεκριμένα θέματα και ερωτήματα. Αναφερθήκατε στο έλλειμμα της ζήτησης. Δεν αναφερθήκατε όμως στο έλλειμμα επενδύσεων που συμβαδίζει με το έλλειμμα της ζήτησης. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, όλοι οι οικονομολόγοι συμφωνούν ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης σταμάτησαν οι επενδύσεις και οι ιδιωτικές και οι δημόσιες. Και μερικές χώρες δεν έκαναν επενδύσεις για να αποφύγουν ε, ε, θετικά εξωτερικά στοιχεία. Έχει νόημα ε, ένα τμήμα του ελλείμματος της ζήτησης να το αναλάβει μια Ευρωπαϊκή Ένωση με πραγματική δημοσιονομική ικανότητα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, πιστεύετε, είναι λογικό κάτι τέτοιο ή εφικτό. Ακούσαμε το διοικητή της ε, Ολλανδικής Τράπεζας, Κεντρικής Τράπεζας και χθες ακούσαμε τον Ολλανδό Υπουργό Οικονομικών στην Επιτροπή Τάξε για τις φορολογικές πρακτικές και ακούστηκε ότι θα πρέπει να είναι ουδέτερη από δημοσιονομική άποψη αυτή η δημοσιονομική ικανότητα. Ενώ μιλήσαμε για μια ανταλλαγή κυριαρχίας και δημοσιονομικής ικανότητας και όλοι είπαμε ότι υπάρχουν πολλές εκτιμήσεις αλλά ακούστηκαν και 100 εκατομμύρια μερικές φορές φοροδιαφυγής που χάνουμε. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν με μια δημοσιονομική ικανότητα να καλύψουμε ένα τμήμα αυτό των ζημιών. Σε ό,τι αφορά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Ραγκό. Αλλά μην ξεχνούμε, μας είπατε για το 2-3%, αλλά το 1929 ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός ήταν 2,5% του ΑΕΠ, ενώ 11 χρόνια μετά είναι 15%. Έγινε 15% το ΑΕΠ. Και ήταν ένας ε, πραγματικός ε, ομοσπονδιακός προϋπολογισμός με όλες τις συνέπειες. Και μάλιστα όλη αυτή η διαδικασία και της αύξησης ε, του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού έγινε σε μια περίοδο δυσπραγίας και κρίσης. Μετά το 29 και ένα θέμα που είναι κάπως συναφές με τη δημοσιονομική ικανότητα. Χρόνια ολόκληρα παρατηρούσαμε ότι οι ανισορροπίες μερικές φορές οφείλονται στη μη συμμόρφωση των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τα κριτήρια για τη συγκράτηση του ελλείμματος και την απώλεια της δημοσιονομικής ισορροπίας αυτές οι αποκλήσεις ε, καταγγέλθηκαν ε, ή επιβλήθηκαν κυρώσεις. Όχι, ούτε το ένα έγινε ούτε το άλλο. Ούτε ε, τις καταγγελίες έγιναν, ενώ αντίθετα αναφέρθηκαν ε, τα πλεονάσματα κάποια χώρα και συγκεκριμένα της Γερμανίας. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο δεν είχε νόημα, αλλά δημιουργεί επιπλέον ισορροπίες αυτή η ύπαρξη ταυτόχρονα ελλειμματων και πλεονασμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλου σκιώδε στην αίθουσα, οπότε να δώσουμε και πάλι το λόγο στου εμπειρογνωμονέ μα. Ο κύριο Κερέ. Με συγχωρείτε, ελέγχω βήχα. Δεν είναι το δημοσιονομικό περιθώριο το προβλήμα μου, αλλά το φωνητικό. σε αυτό που είπε ο συμπρόεδρος, ο κ. Σαρτή προηγουμένως, που ανέφερε τα λόγια μου, ότι η ΕΚΤ ξεπέρασε τις θερμοβίτητες της. Όχι, δεν είπα αυτό. Υπάρχει σαφής, παρτίο αρμοδιοτήτων από τη συνθήκη για μας και το ελέγχετε εσείς ήδη. Δεν θα επεκταθώ εδώ. Αυτό που αληθεύει είναι ότι θα ήταν πολύ απλούστερο για μας εάν ήταν αποτελεσματικότερες οι πολιτικές της Ένωσης για τη δημοσιονομική πολιτική πιο συγκεκριμένα και γενικότερα. Αυτό για να αποσύρω και την ευθύνη από τους ώμους μας. Νομίζω λοιπόν ότι συμφωνούμε έτσι κι αλλιώς. Ο κύριος Μόρεσαν ρώτησε ποιες μεταρρυθμίσεις χρειάζονται. Βεβαίως αυτή είναι μια συζήτηση που θα μπορούσε να κρατήσει, αλλά ο κύριος Μαραγκάλ έκανε μια παρατήρηση και για τις επενδύσεις. Μεταρρυθμίσεις λοιπόν που θα οδηγήσουν σε περισσότερες επενδύσεις. Αυτό νομίζω είναι η καλύτερη απάντηση. Σε κάποιες χώρες υπάρχει επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά θα πρέπει απλώς οι επενδυτές να ενθαρρυνθούν. Και είναι και φτηνές ε, οι ε, συνθήκες αγοραπολισίας, οπότε υπάρχουν δυνατότητες επενδυτικές και πηγές κέρδους ενδεχομένως. Αυτό μπορεί να ε, ενισχύσει και τη συλλογικότητα και με φέρνει στην προηγούμενη παρατηρήσή μου αυτή. Βραχυπρόθεσμα μόνο μπορούμε να δούμε τα πράγματα, όχι μακροπρόθεσμα. Ε, θέλουμε επενδύσεις που θα οδηγήσουν σε παραγωγικότητα και υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι ανάλογα με την κάθε χώρα. Και θα συμφωνήσω με τις προηγούμενες παρατηρήσεις περί κόστους Θέλουμε παραγωγικότητα να δημιουργήσουμε, και επενδύσεις για να μειωθεί το κόστος. Βεβαίως και να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα. Και έγινε μια παρατήρηση από τον κύριο Ντεμάζη. για την πάυση της διασύνδεσης του κρατικού χρέους με τον ε, μάλλον τη διασύνδεση των τραπεζών ε, και ε, το κατά πόσο ένα μηχανισμός εξυγίανσης μπορεί να ε, ενισχυθεί χάρη σε αυτό το μηχανισμό. Με κονδύλια της ΕΚΤΑ δεν μπορεί να λειτουργήσει για την ώρα μόνος ο μηχανισμός στήριξης. Θα ήταν δύσκολο ο Ευρωπαϊκό Μηχανικό Στήριξη να χρηματοδοτείται απολύτω και μόνο από την ΕΚΤ, χωρί να υπάρχει καμία χρηματοοικονομική ε, συνεισφορά. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κνότ. Ευχαριστώ. Ξεκινώ λέγοντα ότι συμφωνώ σε πολλά από αυτά που αναφέρατε για την απουσία των επενδύσεων, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων κτλ. Μπορώ να προτείνω, να αντιπροτείνω ότι η χρηματοδότηση ως κόστος δεν αποτέλεσε εμπόδιο μέχρι τώρα για την Ευρωζώνη. Άρα το πρόβλημα δεν ήταν στην απουσία επενδύσεων. Στην ε, στην παραγωγικότητα ήταν στην ανάπτυξη, στην επένδυση, δηλαδή στην απουσία διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Και κάτι ακόμη μπορώ να προσθέσω για τον κύριο Κορέ. Είναι ότι η σύνθεση των μεταρρυθμίσεων χρειάζεται λίγο περισσότερη προσοχή. Πολλές χώρες που έχουν μεταρρυθμίσεις εστιάζουν τι μεταρρυθμίσει του στην αγορά εργασία, αλλά σε ακραίε καταστάσει, Αν μεταρρυθμίσουμε μόνο την ε, αγορά εργασία και όχι και την αγορά προϊόντων ταυτόχρονα. Το μόνο που κάνεις είναι να μεταθέτεις το βάρος από την αγορά εργασίας στην αγορά προϊόντων. Άρα δεν διορθώνεις τίποτα και έμφαση πρέπει να δοθεί επίσης και στις μεταρρυθμίσεις προϊόντων σε πολλές χώρες και επίσης αυτό βελτιώνει και την αποδεξιμότητα των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις θεωρούνται ε, άνωθεν επιβεβλημένες ε, και βλαβερές για τον εργαζόμενο και προς όφελος του κεφαλαίου. Χρειάζεται λοιπόν ένας καλός συνδυασμός μεταρρυθμίσεων, παραγωγικότητα που θα ενισχύεται χάρη στις επενδύσεις και, αυτές, και αυτή με τη σειρά της θα οδηγεί σε νέες επενδύσεις. Για τις ε, μακροοικονομικές ανισορροπίες του πλεόνασμα πιστεύω τρεχουσών συναλλαγών είναι εσωτερική ανισορροπία, άρα οι προσπάθειες ε, δεν πρέπει να αφορούν μόνο τις χώρες που έχουν έλλειμμα. Για την Ισπανία και την Ιρλανδία βεβαίως το πρόβλημα δεν οφειλόταν στην δημοσιονομική υπερσπατάλη αλλά στο, ε, την εκτός ελέγχου κίνηση της αγοράς τραπεζικής και κυρίως και τα θέματα της ε, από διάρθρωσεις που έφερε σχέση με την αγορά κινήτων, εισαγωγή διαφορετικών φόρων ε, ακίνητης περιουσίας κτλ. Αυτή η ανελαστικότητα λοιπόν είναι πολύ σημαντική να κοιτάξουμε. Ίσως η ασφάλεια που χρειάζεται, αυτό το buffer κάτω από το 3% σε περίπτωση που ξεπερνάει κάτι το 3% πρέπει να είναι και πιο υψηλό από ό,τι είχαμε στο παρελθόν προβλέψει. Και επίσης πιστεύω ότι αν κοιτάξει κανείς το σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη μπορεί να ε, εστιάζονται περισσότερο στο 3% σαν το όριο ως στοιχείο ε, ελέγχου, αλλά το κύριο που πρέπει να τονίσουμε το σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη είναι ότι δεν θέλει το όριο 3%. Θέλει να μην υπάρχουν ανισορροπίε, θέλει σημείο ε, ισορροπία. Σημείο κίνηση λοιπόν που θα ήταν καλύτερο από ό,τι αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε. Η φόρη είναι καθαρά πολιτικό ζήτημα και νομίζω δεν πρέπει να το σχολιάσω εγώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ραγκό. Mm. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω γαλλικά. Επιγραμματικά και πάλι. Το θέμα των επενδύσεων στην Ευρωζώνη, κέριο ζήτημα. Και το έλλειμμα στις επενδύσεις είναι μεγάλο πρόβλημα. Όταν αναλύουμε το έλλειμμα των επενδύσεων, διαπιστώνουμε ότι η βασική αιτία είναι το έλλειμμα στη ζήτηση. Και το βλέπουμε σε όλες τις χώρες. Δεν υπάρχουν παραγγελίες, ε, δεν υπάρχει ζήτηση και αυτό επηρεάζει και τις επενδύσεις. Υπάρχει έλλειμμα των επενδύσεων λόγω του έλλειμματος ζήτησης. Από μακροοικονομική άποψη το έλλειμμα επενδύσεων ε, συνδέεται με τη δυναμική των τιμών και το έλλειμμα της ζήτησης και πολλοί τομείς υφίστανται από πληθωριστικές πιέσεις κάτι που δεν δημιουργεί κίνητρα για τις επενδύσεις και υπάρχει και το ζήτημα δεύτερος παράγοντας, η αβεβαιότητα που έχει και μια ευρωπαϊκή διάσταση. Brexit για παράδειγμα, προσφυγικό, προσφυγική κρίση, συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού πλαισίου. Αυτοί οι δύο παράγοντες, ε, έλλειμμα ζήτηση και αβεβαιότητα, αυξανόμενη βεβαιότητα σε ένα περιβάλλον, επηρεάζουν τις επενδύσεις ε, και άρα υπάρχει το έλλειμμα επενδύσεων. Θα πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα, ισχυρό μήνυμα για υπέρ του ευρωπαϊκού οράματο και το ότι έχει μείνει ζωντανό και να φανεί η βούληση, η πολιτική βούληση ότι ε, θέλουμε να βρούμε λύσει. Γιατί μερικέ φορέ ακόμη και η έκφραση τη βούληση μα λείπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα, σημαντικό μηχανισμό, πολύ σημαντικό εργαλείο για τον επιμερισμό των κινδύνων και την διαχείριση των ευρωπαϊκών κρίσεων. Την ευρωπαϊκή διαχείριση των κρίσεων, μάλλον. Καταλαβαίνω αυτό που είπε ο κύριο Κερέ για τη δυνατότητα έκδοσης τίτλων από το ΕΣΕΜ που θα αγοράζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό εντάσσεται στα πλαίσια ενός ρεαλισμού που χαρακτηρίζει οι νομισματικές ενώσεις και άλλων χωρών όπως τον ΙΠΑ ΕΕ ή τον, του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά που στα πλαίσια των συνδικών θα ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Το να συμμετέχει όμω η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρηματοδότηση μακροοικονομικών εργαλείων, αυτό είναι κάτι που γίνεται και σε άλλε νομισματικέ ενώσει, δημοσιονομικέ ενώσει και κυρίω στι ΗΠΑ. Δεν μίλησε για τη δυνατότητα ε, συμπερίληψη του χρυσού κανόνα. Του να αποκλείσουμε δηλαδή τι επενδύσει από τη, τον υπολογισμό του ελλείμματος σε περίπτωση σημαντικής ύφεση, για παράδειγμα, μια χώρα θα μπορεί να αποκλείσει τις επενδύσεις της από τον υπολογισμό του ελλείμματος. Και γιατί λέμε μόνο σε περίπτωση κρίσης. Για δύο λόγους. Πρώτον, είναι δύσκολο να σκεφτούμε ότι οι δημόσιες επενδύσεις, οι κρατικές επενδύσεις ε, είναι αντικυκλικές. Όταν βλέπουμε το χρόνο εφαρμογής, βλέπει εφαρμογή του σχεδίου Juncker των δημοσίων επενδύσεων, οι δημόσιες επενδύσεις που έχουν σημαντική λειτουργία σύγκληση στην Ευρωζώνη ε, δεν έχουν αντικυκλική λειτουργία. Το να μην σταματήσουμε όμως τις κρατικές επενδύσεις σε μια σημαντική θέση, αυτό είναι το επιθυμητό και το εφεκτό το ευκταίο. Γιατί μερικέ φορέ για τι κρατικέ επενδύσει οι δημόσιε επενδύσει χρειάζονται μακροχρόνιοι ορίζοντε. Γι' αυτό από μακροοικονομική άποψη είναι σημαντικό. Οπότε θα πρέπει να μειώνουμε τις επενδύσεις σε, σε περίοδους κρίσης. Το να τις αποκλείσουμε όμως σε περίοδο κρίσης από τον υπολογισμό του ελλείμματος είναι πολύ σημαντικό και ευκταίο. Σήμερα οι επενδύσεις έχουν και μία πολύ απτή συνιστόσα, τη χρηματοδότηση των υποδομών. Βέβαια, τι επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό, στο εκπαιδευτικό σύστημα, στο σύστημα υγείας ε, δεν είναι ποσοτικοποιήσιμες. Αλλά και αυτές θα πρέπει να τις διαφυλάξουμε σε περίοδους ύφεση. Και μερικέ φορέ στου κανόνε προσαρμογή δίνεται περισσότερη έμφαση στι υποδομέ βάρο των επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό. Θα πρέπει όμω να κρατήσουμε και αυτέ τι επενδύσει, γιατί είναι σημαντικέ και επενδύσει στο ανθρώπινο κεφάλαιο για να υλοποιήσουμε την επιθυμητή σύγκληση. Δεν θα πρέπει λοιπόν να προσανατολίζουμε υπερβολικά το χρήσιμο κανόνα στι υποδομέ, αγνοώντα, αμελώντα το ανθρώπινο δυναμικό. Ε, δεν είναι ε, αντικυκλικέ οι επενδύσει στι υποδομέ και γι' αυτό ακριβώ ε, σκεφτήκαμε το χρυσό κανόνα και συμφωνώ ότι δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί και ο προκυκλικός χαρακτήρας σε εθνικό επίπεδο. Τώρα για τις υπόλοιπες λειτουργίες δεν θα προλάβω να απαντήσω στον κύριο Αρτουή. Μίλησε για την ασφάλιση ανεργίας γιατί έχει κάποιο χαρακτήρα σύγκλησης προς τα πάνω της αγοράς εργασίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, ενεργειακή μετάβαση και την δημιουργία μιας ε, ε, στιβαρής ενεργειακής πολιτικής, χρειαζόμαστε επενδύσεις που θα, που θα χρηματοδοτούν το κοινό συμφέρον και δικαιολογεί και αυτό το ενεργειακό ζήτημα την ύπαρξη ενός κοινοτικού προϋπολογισμού. Ευχαριστώ. Τελικό σχόλιο υπάρχει αυτός ο κανόνας γιατί με κάτω από το 1,5% κενό παραγωγικότητας προληπτικά μόνο μπορεί να μην υπολογιστεί το έλλειμμα συγχρηματοδότησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανεπαρκές μένα αλλά πάντως περί αυτού πρόκειται και έχει μόνο προληπτικό χαρακτήρα όπως είπα και όχι διορθωτικό. Για να δούμε λίγο αν ενδιαφέρεται κανείς να στήσει επιπλέον το λόγο με μια διαδικασία catch the Ποιος θέλει. Ζαν, βλέπω ότι τρώγεσαι, τρεις. Ναι, μία συμπληρωματική για τον κύριο Ρακό. Στην επένδυση σχετική με την ζήτηση. Δεν νομίζετε ότι σχετίζονται οι επενδύσεις με το περιβάλλον που επιτρέπει την ε, ε, αποδοτικότητα, όπου δηλαδή δεν υπάρχει αποδοτικότητα δεν μπορούν να γίνονται και επενδύσεις. Και δεύτερη παρατήρηση, η ενιαία αγορά είναι πολύ κατακαιρματισμένη ακόμα. Άρα χρειάζεται ο επενδυτής και δεδομένου ότι χρειάζεται ο επενδυτής προβλεψιμότητα και ξέρει ότι δεν θα μπορέσουν να κηρυθούν ε, οι τροχοί αφού είναι τόσο κατακαιρματισμένη η αγορά. Ένα αναμονή λοιπόν ε, λύσεων που μπορούν να δοθούν ε, αργότερα δεν κάνει τίποτα. Τηλεπικοινωνίες. 28 διαφορετικές αρχές ρυθμιστικές υπάρχουν και πολλοί άλλοι τέτοιοι τομείς. Άρα καλό είναι να κάνουμε έκκληση για επενδύσεις. Αλλά όσο δεν έχουμε τακτοποιήσει την εσωτερική αγορά και όσο δεν έχουμε αναιρέσει αυτή την ε, κατακαιρματισμένη εικόνα για να φέρουμε τις αγορές προς μια σύγκληση, οι πολιτικές ε, και οι επενδύσεις ε, δεν, θα έρχονται. Εγώ λοιπόν σχετικοποιώ αυτό το συσχετισμό με τη ζήτηση, γιατί απαιτείται η πλήρωση κανόνων, προϋποθέσεων που δεν καλύπτονται αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ, Ελίζα. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Απλώς να καταλάβω την άποψη του κυρίου Κερέκη, λέω, όσο την έκτα. Πώς να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του κατοικού χρέους είναι ένα ζήτημα που διαρκώς επανέρχεται. Η Τραπεζική Ένωση είχε να κάνει με αυτό και με πολλά άλλα βέβαια. Και είναι ένας από τους μηχανισμούς για την ε, διαχείριση του κινδύνου. Σκέφτομαι το ενιαίο ε, βιβλίο κανόνων, τον ενιαίο επιπληκτικό μηχανισμό, την ενιαία εξυγίανση και αναχρηματοδότηση. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια σταθεροποίηση από το στοιχείο της Ευρωζώνης προκειμένου να αναχαιτήσουμε, να, να αντιμετωπίσουμε τους άλλους κινδύνους. Πώς βλέπετε αυτό το συσχετισμό. Νομίζω ο κύριος Νότεν μερή το απάντησε, οπότε όποιος θέλει απάντηση, απαντήσει, αλλά ήθελα να καταλάβω ιδίως την άποψη της ΕΚΤ σχετικά. Περβάνς. Εκτός μικροφώνου. Πολύ σύντομη ερώτηση, γιατί την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια τροπολογία στην Ολομέλεια για το πώς να χρησιμοποιήσουμε στο μέγιστο τα ωφέλη από την ΕΚΤ. Νομίζω λοιπόν ότι εφόσον εδώ έχουμε ένα κεντρικό τραπεζίτη, καλό θα ήταν να μπορέσει να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Η πρόταση θα συζητηθεί και αλλού, οπότε καλό θα ήταν να υποφεληθούμε τις παρουσίες του κυρίου Κερέ για να το σχολιάσει. Παρακαλούμε κύριε Κουρέ. Και πάλι με συγχωρείτε, Θα κάνω το καλύτερο μπορώ. Με συγχωρείτε αν υπάρχουν δυσκολίε και οι ιδιαίτερα συγγνώμη για του διερμηνεί που θα είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσουν. Πρώτα απ' όλα για την ερώτηση τη κυρία Μπερέσου. Τι να κάνουμε με το κέρδο μα. Και με τα κέρδη γενικώ τη τράπεζα. Είναι κάτι που το ορίζει ο εσωτερικό κανονισμό τη ΕΚΤ. Ήδη ταπανώνται διανέμονται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες και μετά από εκεί αναδιανέμονται ανάλογα με τις δικές τους διευθετήσεις. Πάντως στο δικό τους ταμείο πηγαίνουν τα κέρδη και κάθε αλλαγή σε αυτό το σύστημα θα πετούσε και αλλαγή μέσω της συνθήκης. Δεν αποφασίζουμε εμείς τι κάνουμε με αυτά τα χρήματα. Δεύτερον, για την ερώτηση της κυρίας Φερέιρα για το κρατικό χρέος και την Τραπεζική Ένωση. Η συζήτηση έχει φίλη. ως μια κίνηση παράλληλη για το ενιαίο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων και την αναχέτηση κινδύνου για τις τράπεζες. Είναι λογικό, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι οι τράπεζες δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο του, τους κινδύνους των ομολόγων. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες έκθεσης των τραπεζών. Είναι η ποιότητα των κεφαλαίων, είναι τα είδη των δανείων που έχουν. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε όλες τις διαστάσεις της Τραπεζικής Ένωσης σε αυτή την περίπτωση. Και επίσης για τις εκθέσεις των ε, κρατών ε, μέσω του χρέους η δημοσιονομική δυνατότητα μας δείχνει ποιες είναι οι υπόλοιπε παράμετροι. Δεν μπορούμε μονομερός να απαιτούμε ε, να καλύψουμε τα προβλήματα όλα με την συνολική εγγύηση των καταθέσεων και τις κρατικές εκθέσεις ή την έκδοση ομολόγων. Όπως είπα προηγουμένως, έχουμε την αίσθηση ότι θα έπρεπε να υπάρξει κίνηση προς τον περιορισμό της έκθεσης των τραπεζών στο κρατικό χρέος, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει με τρόπο συνετό. και ε, σε, ε, με τρόπο συνεκτικό σε σχέση με όσα γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Απέχουμε πολύ από αυτό ακόμα. Τέλο, εάν επιτρέπετε Πρόεδρε, να επανέλθω σε αυτό που είπε η συνάδελφος για την αβεβαιότητα. Υπάρχει πολλή αβεβαιότητα, όπως είπε ο κ. Ραγό, ε, και στην δική οικονομία και στην διεθνή. Όχι μόνο λοιπόν πολιτική αβεβαιότητα, αλλά Υπάρχει βεβαιότητα για το μέλλον της νομισματικής ένωσης, για τους μηχανισμούς που έχουμε για να απορροφήσουμε τους τριγμούς και τα πλήγματα κατά της νομισματικής ένωσης και τους, τις επενδύσεις που θα στηρίξουν την Ευρωζώνη. Μιλάμε για την πεμπτουσία της έκθεσης των πέντε προέδρων. Θα έλεγα λοιπόν αυτό να μας εμπνεύσει. Εάν μπορούσαμε να εξηγήσουμε με τρόπο έβλητο στους Ευρωπαίους πολίτες ποιο δρόμο, σε ποιο δρόμο θα βαδίσουμε Ω Οικονομική και Νομισματική Ένωση για τα επόμενα 5-10 χρόνια, τότε θα του ανακουφίζαμε αρκετά. Η αβεβαιότητα αυτή μπορεί να διαλυόταν σε μεγάλο βαθμό και να συνεισφέραμε στην ανάπτυξη. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που αυτή η συζήτηση είναι τόσο κέρια. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλε συγκεκριμένε ερωτήσεις. Αλλά αν θέλετε εσείς κάτι. Ναι, πολύ ευχαριστώ. Για να συμφωνήσω με τα όσα είπε ο για να μην δοθεί και η εντύπωση ότι υποστηρίζει έναν υπερβολικά αφελή και ινσιανισμό για τις επενδύσεις και αυτό σχετίζεται ασφαλώς με τη θετική δυναμική της Ισπανίας αυτή τη στιγμή. Βράχει πρόθεσμα, πολύ βράχει πρόθεσμα η ζήτηση στην πενταετία. Και μετά πάμε στα 7-8 χρόνια έχουμε στον ορίζοντα τη σύγκληση και την απόδοση, την αποδοτικότητα ανατομέα και αυτό νομίζω είναι χαρακτηριστικό. Ε, βάζω λοιπόν μπροστά τη ζήτηση ως προοπτική σταθεροποίηση και αυτή τη στιγμή ελλείμματος σε ευρωπαϊκές επενδύσεις αν η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα συνεχιστούν, να συνεχίσουν να είναι ελληματικές, θα έχουμε πρόβλημα μακροπρόθεσμο και διαστρωτικό. Αλλά αυτή τη στιγμή μπορούμε να δώσουμε ως επιχείρημα το έλλειμμα σε επενδύσεις για να εξηγήσουμε τις αδυναμίες της ζήτησης. Και σταματώ γιατί υπάρχουν διάφορες ε, αβεβαιότητες, ε, κύριε Κύριε, σωστά είπατε, υπάρχουν αβεβαιότητες και κυρίως σε σχέση με το ελληνικό χρέος και τα, ε, τις πιέσεις. Για μείωση του ελληνικού χρέους κατά τρόπο αξιόπιστο, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ε, όλοι ξέρουν ότι θα συμβεί, θα υπάρξει μια πολιτική σύγκληση για να προχωρήσει το, ευρωπαϊκό, το πολιτικό εγχείρημα της Ευρωζώνης. Καλώς θέλετε εσείς κύριε Κνότ να πείτε κάτι. Ναι. Ήδη είπα τη γνώμη μου για το κρατικό χρέος σας, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι εάν υπάρχει ένας ε, δημοσιονομικός τομέας και θέλουμε να τον εξηγιάνουμε κύρια αρχή, θα πρέπει να είναι ότι ο κίνδυνος πρέπει να τιμολογείται σωστά. Αντίστροφα, η άλλη του νομίσματος είναι ότι εάν ε, υπό τιμολογείται ο κίνδυνος σε διάφορες περιοχές που μπορεί να συμβεί αυτό στον κόσμο, τότε υπάρχει ε, πολύ υψηλή ανάληψη κινδύνου, ε, ακραία ανάληψη κινδύνου και δεν πρέπει η τραπεζική ε, ε να χρησιμοποιούνται κατά αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να υπάρχει σωστή τιμολόγηση του κινδύνου και όπως έχουμε μάθει και από την κρίση, το κρατικό χρέος δεν είναι στο πυρόβλητο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι δεν είναι ασφαλές το κρατικό χρέος πλέον και πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη μακροχρόνιες περίοδους προσαρμογής και ειδικά για τώρα, για να ξεφύγουμε από την κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα, να φτάσουμε σε μια ορθολογική κατανομή πόρων. Στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ που μας τα είπατε και αυτά. Να δώσω σύντομα το λόγο στον κύριο Μπέγκε για μια σύντομη... Μάλλον πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μπέγκε θα ήθελα σύντομα να κάνω μια ε, τεχνικού χαρακτήρα παρατήρηση. Υπάρχει το άρθρο 30, 30 παράγραφος 4 του καταστατιστικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζας που μιλάει για την αναθεώρηση μια δίκη ε, ε, αναθεώρηση που θα μπορούσε να προχωρήσει κατόπιν αιτήματο τη ίδια τη ΕΚΤ. Επομένω, αλλά δεν είσαστε τελείω τελείω αδέκαστοι, αμερόληπτοι και ουδέτεροι ω προ τι συνθήκε. Αντίθετο, έχετε και δικαίωμα πρωτοβουλία. Άρα μπορείτε να σχολιάζετε βεβαίω, αλλά καταλαβαίνουμε ότι σήμερα δεν θέλετε να το πράξετε. Προσπαθώ να αντισταθώ στον πειρασμό, αλλά δεν τα καταφέρνω. σε σχέση με την τιμολόγηση του κρατικού χρέους. Βεβαίως έχετε δίκιο, αλλά, αλλά με ένα πιο περιορισμένο κρατικό χρέος πώς μπορεί ε, να μην καταρρεύσει το σύστημα γιατί εάν υπάρξει στάση πληρωμών σε κρατικό επίπεδο και με 25% και με 35% οι τράπεζες πρόβλημα θα έχουν. Μην λέμε λοιπόν ότι μικρότερη έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε μη πρόβλημα, δεν το έχουμε λύσει. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό της Ευρωζώνης. η σύμβαση της Βασιλείας είναι ο τρόπος να λυθούν όλα αυτά και πρέπει να μετατραπεί το πρόβλημα σε διαχείριση κινδύνου, από διαχείριση κινδύνου σε ανακοίνωση κινδύνου. Πράγμα το οποίο ξέρουμε ότι οι αγορές δεν μπορούν να αντέξουν διαφορετικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και για να πω δύο λογάκια συμπερισματικά. για το έγγραφο εργασία και τους ε, ομιλητές μας. ευχαριστούμε θερμά, μας ε, έδωσαν τα φώτα τους και σε εμά και στους ε, συνεργάτες μας για τα διάφορα ζητήματα που και επιστημονικά αλλά και πολιτικά έπρεπε να συζητήσουμε. Είχα μια εκδήλωση στην εκλογική μου περιφέρεια πρόσφατα και ε, είπα ότι εγώ ως χριστιανοδημοκράτης Γερμανός ανέλαβα μαζί με μια καλύδα σοσιαλίστρια μια πρωτοβουλία αυτού του τύπου όπως σημερινή ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά τη Ευρωζώνη. Είδα τα μάτια των ανθρώπων να μεγαλώνουν και με κοιτάνε με έκπληξη και μου λένε λέει, τώρα γιατί πράγματα συζητήσετε. Ε, και του εξήγησε ότι κοιτάμε για μια κοινότητα ευρωπαϊκή που θα λύνει τα προβλήματα για τον πολίτη. Ταυτόχρονα με υπευθυνότητα ώστε να μην λησμονούμε που πρέπει να τίνει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να διδασκόμεθα από τις κρίσεις και να καταλάβουμε ότι ο κόσμος συνεχίζει να γυρίζει και δεν μας περιμένει από τις τοποθετήσει, από τις αντιδράσεις, διαπιστώνω ότι βρισκόμαστε μόνο στις αρχές της δουλειάς που έχουμε αναλάβει. Αλλά και με τις ε, εκθέσεις μας που θα πάνε στην ε, ε, Ολομέλη αλλά και πιο πριν στις επιτροπές μας θα έχουμε μια έκθεση πρωτοβουλία που θα διατυπώνει ξεκάθαρα τη θέση του Κοινοβουλίου και που θα καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλάβουν υπεύθυνη στάση και συντονισμό για τον Ευρωπαίο πολίτη. Όχι κατακαιρματισμένο, όπως δυστυχώς έχουμε δει τόσο καιρό. Η δημοσιονομική ικανότητα βέβαια δεν μπορεί να αποτελέσει διέξοδο όταν κάποιος δεν κάνει τη δουλειά του στα εσωτερικά του δημοσιονομικά και συμφωνώ ότι δεν είναι η κατάσταση των επενδύσεων αυτή η οποία εμποδίζει αυτή τη στιγμή Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι αν έχει κάνει κάνει επενδύσει πριν από 40 χρόνια ε, και πόσο περισσότερο θα πληρώσει από αυτό που θέλει να κάνει τώρα, αλλά εάν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις επενδύσεις και αν έχουμε επιλογές πιο στοχευμένες και εδώ θα βάλω και τη δική μου ιδιαίτερη πατρίδα βέβαια στο σχέδιο που θα λύνουν μακροπρόθεσμα τα προβλήματα και τις απασχόλησης. Και βέβαια συστάσεις ανακράτος, υπευθυνότητα, ευθύνη, έλεγχος, λογοδοσία, όλα αυτά είναι αισθήματα τα οποία πρέπει να βρουν απάντηση και μερικά από αυτά τα οποία μπορούμε να πράξουμε, όπως υπόθηκε, είναι δυνατόν να υλοποιηθούν και χωρίς αναθεώρηση νοτικών, αλλά υπάρχουν κάποια άλλα σημεία όπου ίσως θα πρέπει να λάβουμε την απόφαση για αναθεώρηση των συνθήκων που φυσικά ξέρουμε όλοι ότι θα κρατήσουν πολύ περισσότερο χρόνο, που θα κρατήσει πολύ περισσότερο χρόνο, αλλά ίσως έτσι μπορούμε να δώσουμε ακροπρόθεσμες απαντήσεις στη προβλήματα της Ευρωζώνης, στη σταθεροποίηση, αυτό τελικά το οποίο δηλαδή περιμένει από εμά ο πολίτης, από εμά ε, ε, ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εισαγωγική μας κουβέντα. Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας για την παρουσία τους και καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστώ.